Ja, ich glaube, wir können langsam anfangen. Wir haben Κυρίε και κύριοι, καλημέρα σα. Σήμερα θα προβούμε σε ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Μάρτσιν Κόρατσεκ, πρώην Υπουργό τη Πολωνική Κυβερνήσεω και τώρα πληρεξούσιο τη Πολωνική Κυβέρνηση για την κλιματική πολιτική. Μάλλον είναι και τώρα ακόμη Υπουργό Περιβάλλοντο Πολωνίας. Τον συναντήσαμε στη Βαρσοβία για τη 19η ε, διάσκεψη για το κλίμα. Είχαμε συζητήσει και με τον κύριο Χιντεκάρτ. Και τώρα θα ακούσουμε από τον ίδιο τον Υπουργό τα αποτελέσματα, την ε, σύνοψη και θα έχουμε και την ευκαιρία να συζητήσουμε διάφορα ζητήματα με τους συναδέλφους. Χωρίς άλλη χρονοτριβή λοιπόν, δίνω το λόγο στον πληρεξούσιο της πολωνικής κυβέρνησης για την κλιματική πολιτική, κύριο Μάρτσιν Κόρολεκ. Έχετε το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. E, Ευχαριστώ πολύ. Όσον αφορά τα αποτελέσματα της διάσκεψης στη Βασοβία, θα ήθελα να εστιαστώ σε δύο πτυχές. Σε δύο είδη αποτελεσμάτων από τη διάσκεψη. Πρώτη πτυχή καταφέραμε να συμφωνήσουμε να λάβουμε από κοινού διάφορες αποφάσεις, να συμφωνήσουμε σε διάφορα συμπεράσματα. Και μιλάμε για αρκετές ε, δεκάδες ε, συμπεράσματα και αποφάσεις. Οι πιο σημαντικές από τις οποίες είναι οι εξής πέντε. Πρώτον, μια απόφαση για την ατζέντα του Ντέρμπαν. Δεύτερον, μια απόφαση για το μηχανισμό απολύων Τρίτον, ένα πακέτο 7 αποφάσεων ε, για τη χρηματοδότηση της κλιματικής πολιτικής. Τέταρτον, υποβολή αναφορών και παρακολούθηση των εκπομπών. Και πέντον, Επτά περίπου αποφάσεις για τη δασοκομεία, για την ε, δασοκομική πολιτική στις τροπικές χώρες. Επιτρέψαμε να επεκταθώ λίγο σε αυτές τις ε, πέντε μίζωνες αποφάσεις. Πρώτον, η πλατφόρμα του Ντέρμπαν καταφέραμε να καταλήξουμε σε έναν οδικό χάρτη και εν ώψη της ε, διάσκεψης των Παρισίων θα γνωρίζουμε τι θα συμβεί και πότε μέσα στα επόμενα δύο χρόνια. Υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα. Έτσι λοιπόν ε, η διάσκεψη του Παρισιού ελπίζουμε ότι θα μπορέσει να λήξει με επιτυχία. Όλοι γνωρίζουμε ότι το πρώτο σχέδιο, το προσχέδιο απόφασης, το πρώτο σχέδιο απόφασης θα υποβληθεί στα μέρη ακριβώς πριν από τη διάσκεψη στη Λίμα το Δεκέμβριο του επόμενου έτους. Στη Λίμα τα μέρη θα συζητήσουν και θα συμφωνήσουν για το πώς θα παρουσιάσουν τις, ε, τις συνεισφορές τους, ε, τη συμβολή τους στη νέα συμφωνία. Οι συμβολές αυτές θα πρέπει να παρουσιαστούν στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2015. Επίσης γνωρίζουμε ότι το Μάιο του 2015 θα πρέπει διανεμηθεί το σχέδιο συμφωνίας ε, σε όλες τις επίσημες γλώσσες ε, της διάσκεψης τη σύμβαση, συγγνώμη, πριν από, έξι μήνες πριν από τη διάσκεψη στο Παρίσι. Ο δικός χάρτης λοιπόν συμφωνήθηκε. Συμφωνήθηκε δηλαδή το χρονοδιάγραμμα από σήμερα μέχρι τη διάσκεψη του Παρισιού και η, η απόφαση στη Βαρσοβία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συμμορφώνεται απόλυτα με την απόφαση που ελήφθη πριν από δύο χρόνια από τα μέρη του διάσκεψης του Ντέρμπαν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό ότι οι αποφάσεις ε, του Ντέρμπαν, της Λίμα, της Βαρσοβίας και εν τέλει του Παρισιού θα είναι απολύτως συμβατές. Ώστε κανείς να μην μπορεί να ισχυριστεί ότι η διαδικασία δεν έχει νομιμότητα ή δεν τήρει τις αρχικές αποφάσεις που ληφθήκαν στον Τέρμπαν. Οι υπόλοιπε τέσσερις αποφάσεις, η δεν τηρει τις αρχικες αποφασεις που ληφθηκαν στον τερμπαν οι υπολοιπες τεσσερις αποφασεις η αποφαση για το μηχανισμό απολειών και ζημιών ε, βασίστηκε σε πολύ δύσκολες διαπραγματεύσεις. Ειδικότερα οι νησιωτικές χώρες και οι αναπτυσσόμενες χώρες ε, προσδοκούσαν εδώ και πολλά χρόνια για αυτή την απόφαση. Ε, οι αρχές της διάσκεψης χαρακτηρίστηκαν από τα τραγικά γεγονότα στις Φιλιππίνες και στις υπόλοιπες χώρες της περιοχής. Ε, και το ότι συμφωνήθηκε ο μηχανισμός ε, απολειών και ζημιών, ε, αυτή η συμφωνία είναι ιστορική σημασία. Έτσι, σήμερα μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση για τους μηχανισμούς αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών. Το τρίτο σημείο, τρίτη πτυχή που ανέφερα, πολύ σημαντική, πολύ ευαίσθητη, ήταν το ζήτημα της χρηματοδότησης της κλιματικής ε, πολιτικής. Και εδώ από τις επτά αποφάσεις θα ήθελα να εστιαστώ στις δύο, που βασίστηκαν σε πολύ δύσκολες διαπραγματεύσεις. Η πρώτη αφορούσε τις επιχειρησιακές πτυχές του κλιματικού ταμείου και η απόφαση για τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της κλιματικής πολιτικής. Και οι δύο αποφάσεις ήταν πολύ δύσκολες, πολύ ευαίσθητα θέματα, αλλά καταφέραμε να καταλήξουμε συμφωνία για αυτά τα σημεία. Η τέταρτη πτυχή, πολύ σημαντική, παρότι όπως χειρίζονται ορισμένοι πολυτεχνικοί, το ζήτημα της υποβολής εκθέσεων και μέτρησης της μείωσης, ε, μετρής δηλαδή των μειώσεων από τα κράτη-μέλη. Είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, ειδικότερα επειδή ειδικότερα επειδή ετοιμαζόμαστε να ε, επειδή συμφωνούμε για κάτι δεσμευτικό για όλα τα κράτη-μέλη. Ε, και τέλος η συζήτηση για τη δασοκομεία, η συμφωνία για τη δασοκομεία, ε, τη δασοκομεία στα τροπικά δάση. Μια βιώσιμη ατζέντα για τα τροπικά δάση. Αυτή είναι, αυτό είναι το τεχνικό κομμάτι της διάσκεψης. Επίσης, ε, ελήφθησαν ε, μεγάλο πλήθος άλλων αποφάσεων. Αλλά θα ήθελα να επισημάνω και άλλη μια πτυχή, μια άλλη διάσταση, εξίσου σημαντική. Ε, αυτής εξ αρχής, μία από τις φιλοδοξίες ήταν να επανακτήσουμε την εμπιστοσύνη μας στη διαδικασία. και να επανακαθιερώσουμε τις αρχές της διαφάνειας και γενικά της οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Όπως φαίνεται, αυτό το τεχνοκρατικό νόημα ή το αποτέλεσμα μάλλον των αποφάσεων μιλάει από μόνο του. Αποδείξαμε ότι ακόμα και σε πολύ δύσκολες εποχές και υπό δύσκολες περιστάσεις είναι δυνατή η επίτευξη συμφωνίας. Τώρα το ζήτημα της οικοδόμησης εμπιστοσύνης πραγματοποίησης της διάσκεψης είναι κάτι άλλο. εμπνευστήκαμε από τις εργασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και για πρώτη φορά στην ιστορία παρουσιάσαμε το θεσμό του τρίου προεδρίων Πολωνικής, Περουβιανής και Γαλλικής. Τρία προεδρίων λοιπόν, Πολωνίας, Γαλλίας και Περού όλες οι συναντήσεις με τη γραμματεία οι οποίες συνήθως λαμβάνουν χώρα καθημερινά ή μάλιστα και περισσότερες από μία φορά, φορά την μέρα σε όλες τις συναντήσεις καλέσαμε τις μελλοντικέ δύο προεδρίες την Περουβιανή και την Γαλλική να συμμετάσχουν ενεργά στις συναντήσεις Καλές, καλούσαμε επίσης τις ε, δύο αυτές προεδρίες ε, σε όλες τις συναντήσεις του Προεδρείου. Στις συναντήσεις γεωγραφικών ομάδων και γραμματείας, ε, αυτές οι συναντήσεις λαμβάνουν χώρο δύο φορές την εβδομάδα και έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν απολογισμό της προόδου των ε, υποεξέλιξη διαπραγματεύσεων. Όλες οι γεωγραφικές ομάδες λοιπόν εκπροσωπούνται σε αυτές τις συναντήσεις και σε όλες αυτές τις συναντήσεις παρέστησαν και εκπρόσωποι των δύο επερχόμενων προεδριών. Επίσης αποφασίσαμε να καλέσουμε μια σειρά υπουργών να συμμετάσχουν στη διαδικασία. Και αυτό είναι μια καινοτομία. Για παράδειγμα, όσον αφορά τη χρηματοδότηση των κλιματικών πολιτικών και του μηχανισμού απολειών και ζημιών και τις διαπραγματεύσεις ε, της συμφωνίας μας βοήθησαν ε, πολλοί υπουργοί. Για παράδειγμα, το ζήτημα της χρηματοδότησης ε, υπήρχε υπουργό Λίντεγκαρντ από τη Δανία και ο Υπουργός Κίβανουφ από την Ουγκάντα για τις ζημίες και τις απώλειες ε, μας βοήθησαν ε, οι Υπουργοί ε, Λένα Εκ της Σουηδίας πρώην Ευρωβουλευτής και η Εντνα Μόλενα από την Νότια Αφρικανική Δημοκρατία. Τώρα, όσον αφορά τη νέα συμφωνία, μας βοήθησαν ε, ο Έντιμ Κράσερ από την Ισλανδία και ο κύριος Μπαλακρίσνα από την Σιγκαπούρη. Πιστεύω ε, το γεγονό αυτό ότι συμμετείχαν ε, μια σειρά υπουργών στις ε, διαβουλεύσεις μας και μάλιστα και αρκετοί Ευρωπαίοι υπουργοί και ο Φιλανδός υπουργό ήταν που διευθύνει τη συζήτηση για το πώς τα δάση και η δασική πολιτική συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών. Και πιστεύω ότι η αρρωγή τόσων πολλών υπουργών περιβάλλοντος ε, συνέβαλε στα καλά αποτελέσματα, στο μεγάλο πλήθος αποφάσεων που λήφθησαν. Αλλά συνέβαλαν επίσης και στο γεγονός ότι καταφέραμε να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη στη διαδικασία παράγοντας τόσο σημαντικός σε αυτή την περίοδο πριν από το τελικό φινάλε που θα λάβει χώρα στο Παρέσι σε δύο χρόνια. Διότι μόνο εφόσον υπάρχει εμπιστοσύνη από τους ε, διάφορους υπουργού και τους διαπραγματευτές εμπιστοσύνη στο ότι η διαδικασία ε, είναι χωρίς αποκλεισμούς, είναι διαφανής. Ε, μόνο έτσι θα μπορέσει να καταστεί δυνατή μια συμφωνία στο Παρίσι. Είμαστε πεπισμένοι ότι έτσι και θα συμβεί στο Παρίσι. Αυτό θα συμβεί, θα καταλήξουμε στη συμφωνία. Θα κλείσω εδώ και ευχαρίστω να απαντήσω τις ερωτήσεις και να ακούσω τα σχολεία σας, εφόσον υπάρχουν. Σα ευχαριστώ κύριε Κόρολεκ. Αγαπητοί συνάδελφοι, δύο. Έχω το λόγο, Εστρέλα. Γκίρεκ. Ξεκινάω με τον κύριο Άγιχαουτ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Και ευχαριστώ καταρχάς τον κύριο Κόρολετς. Έχουμε τις διαφορές μας καμιά φορά. τι απόψεις, ανταλλαγές, tweets, πολύ ενδιαφέρουσες και ευχαριστώ πολύ τον κύριο Κόρολες και θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω για τα καταληκτικά λόγια από την, από την ε, ε, διάσκεψη της ε, Βαρσοβίας το ότι κάνατε την παρέμβαση αυτή το, το Σάββατο παρά τις διαφορές και τα προβλήματα ήταν πάρα πολύ σημαντικό και ήθελα να το δηλώσω και από εδώ. Μία ερώτηση γιατί η Βαρσοβία ήταν ε, μια διάσκεψη που είχε δυσκολίες, δεν ήταν καθόλου εύκολα τα ζητήματα. Πολλές χώρες και στο διεθνές πεδίο δεν ε, συνεργάστηκαν όπως τα περιμέναμε. Για να είμαστε όμως κάπως πιο σαφείς ως προς την κατάσταση, μπορείτε να μου εξηγήνετε τι γίνεται σε σχέση με τον Υπουργικό σας θόκο, τι συνέβη μετά την διάσκεψη το κλίμα και από εδώ και μπρος τι γίνεται. Τι συνέπειες δηλαδή θα φέρει αυτή, εφόσον είσαστε ακόμη από ό,τι βλέπω αρμόδιος για την κλιματική πολιτική, θα ήθελα να μάθω πιο πολλές λεπτομέρειες για τι συνέβη εκεί και ποιος ακριβώς θα είναι ο δικός σας ρόλος. Η πιο σημαντική βέβαια, το πιο σημαντικό θέμα συζήτηση είναι ότι τώρα πια που έχουν ε, ε, αποσοβηθεί κάποια από τα προβλήματα που είχαμε ως τις απώλειες και τη ζημία, ε, μπορούμε ίσως με τη χρηματοδότηση, εφόσον προχωρήσουμε συζήτηση από ό,τι τουλάχιστον φαίνεται, και ξαναγυρίσει το θέμα στην ημερήσια διάταξη για το Περού αλλά και για το Παρίσι ελπίζω, ε, μένει οπωσδήποτε να δούμε το θέμα του φίλου πορείας μέχρι το Παρίσι. Ε, πώς μπορεί να προωθήσει το θεματολόγιο αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί βέβαια φαίνεται πως είναι πολύ σημαντικό να έχουμε επαρκείς επιλογές. Και ίσως θα πρέπει και εσείς ε, να μας προτείνετε ιδέες για το πώς μέχρι το 2014 η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να διαμορφώσει τις θέσεις, τις θέσεις της μετά την, ε, με βάση μάλλον και την πλατφόρμα του Durban. Τα άρθρα ε, επί παραδείγματι 5C για τον περιορισμό των εκπομπών 4C για τις ε, χώρες που υπάγονται στη δεύτερη περίοδο δεσμεύσεων της, της, ε, του πρωτοκόλλου του Κιώτο, ε, βασικά ευρωπαϊκές χώρες, δηλαδή όπου ζητείτε να αναπτυχθούν πιο φιλόδοξοι στόχοι. Και επίση ε, θα ήθελα προτάσεις για το 4C, πώ μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να το χειριστεί. Μετά δε την περίοδο 2020 καλούνται τα μέρη να καταθέσουν προτάσεις δράσεως μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2015 εφόσον είναι σε θέση, τουλάχιστον αυτή είναι η διατύπωση, είναι δηλαδή σαφές ότι αυτή η περίοδος, το πρώτο τρίμηνο του 2015, επιλέγεται για να έχουν ε, ε, πραγματοποιηθεί οι εκλογές, οι ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες και άρα να είναι έτοιμες και εκείνες από πλευρά τους να συμπράξουν. Αλλά από το 2014 και μετά η Ευρωπαϊκή Ένωση τους ή άλλως θα πρέπει να φέρει αποτελέσματα πιο απτά για την περίοδο μετά το 2020. Και γι' αυτό θέλω και εσείς ως επικεφαλής βεβαίως της διασκέψεως για την κλιματική αλλαγή πολιτική όπου βλέπετε από πλευρά σας κάποιες κυβερνήσεις και της Ευρωπαϊκής Ενώσης βεβαίως να προβαίνουν σε νέες επιλογές και αλλαγές αλλά και από τη θέση σας ως ε, Πολωνού Υπουργού ε, θα ήθελα να δω τι μπορείτε να προβλέψετε για τις κινήσεις Πολωνίας από εδώ και μπρος και βέβαια για τον προσεχή Μάρτιο και για την Σύνοδο Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετά την απόφαση κόπου για την οποία τόσο πολύ αγωνιστήκατε και εσείς. Θα λοιπόν τις απόψεις σας. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Στρέλα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον Υπουργό για την παρουσία του και για, να τον ευχαριστήσω και για όλες τις πληροφορίες που μας έδωσε. Σε σχέση τώρα με τα αποτελέσματα της διάσκεψης COP19, μας έρχεται η εικόνα του μισοάδιου μισογεμάτου ποτηριού. Το αποτέλεσμα είναι το μισο άδειο για κάποιους διότι δεν επιτέθησαν τα ουσιαστικά και άλλοι το βλέπουν μισογεμάτο. Εν ολίγης υπήρξαν και αρνητικά και θετικά στοιχεία. Νομίζω επ' αυτού θα συμφωνήσουν όλοι. Ως προς τα αρνητικά στοιχεία, θα έλεγα και ορισμένες φορές δεν φαίνονται αρκετά σημαντικές ε, οι λέξεις, αλλά παρόλα αυτά έχουν ένα σημαντικό σημασιολογικό φορτίο. Ε, μιλώντας, μιλώντας λοιπόν για τους ε, συμβιβασμούς, θα μπορούσε κανείς να μιλήσει για υποχώρηση. Αυτό είναι το πρώτο αρνητικό στοιχείο. Επίσης αρνητικό μου φαίνεται το ότι όχι μόνο από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και από πλευράς διαφόρων με, συμβαλωμένων μέρων δεν υπήρξαν αρκετά υψηλές φιλοδοξίες. Ως προς την Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρώ ότι είναι λυπηρό πως δεν παρουσιάστηκε το μέτρο της μείωσης κατά 30% των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα μέχρι το 2020. Αυτό από μόνο του μας λέει πολλά πράγματα διότι έχει συζητηθεί επί μακρόν και εδώ και πάρα πολύ καιρό αυτό το ζήτημα. Βλέπουμε λοιπόν ότι δυσκολευτήκαμε να καταλήξουμε σε μια συνένεση εδώ στο Κοινοβούλιο ακόμη και ε, ε, ε, για αυτό το μέτρο και μόνο. Ως προς τις ίδιες τις αποφάσεις που ελήφθησαν, είναι προφανές ότι είναι προτιμητέο να έχουμε αυτό τον οδικό χάρτη που έχουμε παρά να μην έχουμε κανέναν. Ναι. Αναβάλουμε όλα τα στάδια των διαπραγματεύσεων μέχρι το Παρίσι. Το 2015 παραφορτώνοντας έτσι την ημερήσια διάταξη του 2014. Πιστεύουμε δηλαδή ότι το 2014 θα επαρκέσει χρονικά για να προετοιμάσουμε το θεματολόγιο το 2015. Πώς θα υλοποιηθούν πιστεύετε τα διάφορα στάδια αυτής της πορείας. Και προσθέτω ότι θα ήταν ε, πιο θαραλέο από πλευρά μα να είχαμε ε, προδιαγράψει την πορεία μα μέχρι το 2020 και όχι το 2014. Επανέρχομαι και πάλι στα αρνητικά σημεία, αλλά δεν μιλώ αποκλειστικά πλέον για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι λυπηρό που η Ιαπωνία και ο Καναδάς που σε άλλες κόπ είχαν αρκετά επικοδομητικό ρόλο, όπως στην κόπ του Μόντρεαλ για προφανείς λόγους ε, είχε και υψηλότερη δέσμευση ο Καναδάς, καρκινοβατούν και ο Καναδάς και η Ιαπωνία σε σχέση με την προηγούμενη ΚΟΠ. Λυπηρό και αυτό. Ας περάσω και στις θετικές πλευρές. Ε, το ζήτημα της χρηματοδότησης που είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα μπορέσαμε να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Εγώ θεωρώ θετικό το ότι στον τομέα της χρηματοδότησης ε, αποφασίστηκαν τα περί πρασίνου ταμείου για την ανάπτυξη, ο διεθνής μηχανισμός της Βαρσοβίας όπως τον ε, αποκάλυψαν η μείωση των εκπομπών για την αποψήλωση των δασών 280 δις δολάρια ε, είναι το κονδύλι που τελικά αποφασίστηκε. Θετικό αυτό όμως. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να έχει δραστηριοποιηθεί περισσότερο και θα έπρεπε κυρίως να έχει υψηλότερες φιλοδοξίες. θα έπρεπε να έχουν γίνει περισσότερα βήματα για να προσεγγίσουμε το 2015 ώστε να έχουμε καλύτερες πιθανότητες να συνάψουμε τη συμφωνία το 2015 ή κάποια ε, σημάδια υποχώρησης ε, μας απογοητεύουν, μας αποθαρρύνουν αντί να ε, προχωρούμε, υποχωρούμε ε, Ε, στο δίκτυο κλιματικών επιδόσεων των μηχανικών χωρών η Πορτογαλία είναι στην τρίτη θέση σε σχέση με τις επενδύσεις που έγιναν στον τομέα κυρίως των ανανεώσιμων. Τώρα όμως ε, λόγω της κρίσης, ε, λόγω της τροποποίησης της εθνικής πολιτικής ήδη ακολουθεί λάθος κατεύθυνση, δεν προχωράει. Τέλος. Θα ήθελα να προσθέσω κάτι για τις ε, μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Κάποιες αποφάσισαν ε, να αποχωρήσουν, να ε, μην συμμετάσχουν πλέον στις εργασίες. Υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος που θα αιτιολογούσε μια τόσο ριζοσπαστική αλλαγή ερώτας για τις μικρόν, Ευχαριστούμε κυρία Εστρέλα ο Άνταμ Γκίρικ, τελευταίο ομιλητής και συνέχεια Εσημάνσκι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ. Πόσο δύσκολη ήταν η διάσκεψη. Και αντιλαμβάνομαι ότι οι αναδυόμενες χώρες αλλά και οι χώρες του, κόσμου, του τρίτου κόσμου τα προβλήματα αυτά τα εξετάζουν στο πλαίσιο της κλιματικής δικαιοσύνης. Και αυτό βέβαια προβάλλει μια σειρά από συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ των κρατών Δεν θέλω λοιπόν να αναφερθώ σε αρνητικά ζητήματα κάθε συζήτηση. Κάθε γύρος συζητήσεων θα πρέπει να αξιολογείται με θετικό τρόπο. Και μόνο το γεγονός ότι γίνονται οι συζητήσεις πρέπει να κρυφεί ως ε, θετικό. Υπενθυμίζω ωστόσο στην κυρία Στρελά ότι ο ευρωπαϊκός στόχος παραμένει το 2020-2020. αυτη ήταν και η βάση των συστήσεων μας στη Βαρσοβία. Το πώς θα επιτευχθεί ο στόχος αυτός βέβαια. Γιατί πρέπει να θυμόμαστε ότι αυτοί οι στόχοι εξετάζονται μέσα στον κόσμο, άνα τον κόσμο καλύτερα, στο πνεύμα της κλιματικής δικαιοσύνης. Εκ τούτου δεν μπορούμε να είμαστε υπερβολικά ακραίοι στην παρέμβαση μας, συνδραστικοί στην, στις παρεμβάσεις μας σε ορισμένους τομείς. Χρειάζεται χρήμα, το είπαμε αυτό. Χρειαζόμαστε χρήμα, το είπε και ο Υπουργό. Έχουμε πολλέ φυσικέ καταστροφέ, πολλά επεισόδια, τη μεγάλη καταστροφή στι Φιλιππίνες. Πιο πριν και άλλα προβλήματα. Και η Πορτογαλία, αν δεν απατώ, με έχει γνωρίσει τραγωδίες που έχουν προξενήσει φυσικές καταστροφές. Ας είμαστε προσεκτικοί λοιπόν. Ας είμαστε προσεκτικοί γιατί διατυπώνοντας ε, τις ε, ε φιλοδοξίες μας πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. στη Βαρσοβία καταφέραμε να συμφωνήσουμε στην πολιτική για τα δάση. Αυτό το πέτυχε η Βαρσοβία. Μια πολιτική στον κόσμο ολόκληρο που δεν υπήρχε και αυτό είναι κάτι το πολύ σημαντικό και πρέπει να εξασφαλίσουμε την επιβίωση αυτών των πνευμόνων του πλανήτη μας. Είναι θετικό λοιπόν, πολύ σημαντικό το καταφέραμε. Είναι πολύ σημαντικό το ότι συμφώνησαν τα μέρη και θα ήθελα να συγχαρώ, να επενέσω τους ε, συμβαλωμένους για την επίτευξη αυτή. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω και τον Υπουργό τώρα, γιατί πρέπει να επιτύχουμε αυτό νέο Κιώτο στο Παρίσι και το 2015. Ο στόχος είναι να διαφυλαχθεί η συμφωνία του Κιώτο και με διεύρυνση ενδεχομένω του πεδίου εφαρμογή τη και επέκταση. Αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να δούμε αυτή η συμφωνία του Κιώτο τι, σε τι επίπεδο βρίσκεται, σε τι κατάσταση βρίσκεται. Έχει γίνει σχετική ανάλυση. Η πατρίδα μου παραδείγματι έχει ξεπεράσει κατά πέντε φορές τις προϋποθέσεις της συμφωνίας του Κιώτο. Και ε, θα ήθελα να ρωτήσω λοιπόν τι γίνεται με τέτοιου είδους περιπτώσεις όπου υπάρχει τόσο σημαντική μείωση, δραστική μείωση των εκπομπών. Το συζητήσατε αυτό στη Βαρσοβία, γιατί και στο Παρίσι του έρθει η ώρα για τις ε, εκπομπές. Θα ξεκινήσουμε από το μηδέν. Από το Κιώτο. Ε, το Κιώτο θα είναι η βάση μας. Σας ευχαριστώ θερμά. Ο κύριος Σιμάνσκι έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον Υπουργό μας για την εξαιρετική του συμβουλή και την παρουσίασή του. Θα ήθελα να πω ότι λυπάμαι που δεν είναι πια υπουργό, είναι σημαντικός βέβαια ακόμα, είναι αρμόδιος για το κλίμα, αλλά θα ήθελα να είχατε παραμείνει υπουργό. Θυμάμαι ότι όταν βρισκόσταν εδώ στην Επιτροπή μας ε, την άλλη φορά είχα εντυπωσιαστεί από τις απόψεις και τις ιδέες σας, οι οποίες δεν βρήκαν σύμφωνα όλα τα μέλη. Θα το θυμάστε ότι εκείνη την εποχή είχατε πει πως ένας από τους στόχους της διάσκεψης της Βαρσοβίας δεν ήταν ε, να γίνουν δεσμεύσεις ε, για τελικές αποφάσεις, αλλά επικεντρωθήκατε και επισημάνατε αυτή την πτυχή της Παγκόσμιας Συμφωνίας διότι αυτό θα αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά της όλης αυτής πολιτικής. Αυτή η παγκόσμια συμφωνία είναι πολύ σημαντική. Αυτό είχατε πει. Επίσης είχατε εκφράσει επιφυλάξεις ε, όσον αφορά τις περαιτέρω μειώσεις στην Ευρώπη αν οι υπόλοιπε χώρες δεν ακολουθούν οι υπόλοιπε μεγάλες δυνάμεις. Επίσης είχατε αναφέρει την ε, απελευθέρωση του εμπορίου Είχατε αναφέρει και για το μοτίβο φθηνή ενέργεια ε, εκτό Ευρώπη και ακριβή ενέργεια ε, στην Ευρώπη όσον αφορά τα θέματα δικαιοσύνη, ισότητα, ε, ανταγωνισμού. Αυτά είχατε πει τότε. Όλε οι χώρε. Υποτίθεται ότι πρέπει να πούμε ότι ναι, έχουμε διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης. Ε, έχουμε χώρες που αθέτησαν την υποσχέσή τους και υπάρχουν άλλες ε, χώρες που έχουν διαφορετικά νούμερα. Για παράδειγμα, ένας Κινέζος ε, εκπέμπει δύο τόνους διοξιδίου του άνθρακα αλλά είναι 9 τόνοι στη Γερμανία και στο Λουξεμβούργο είναι 20 αυτοί οι τόνοι. Χρειαζόμαστε λοιπόν κάποια κριτήρια, κάποια σημεία αναφοράς. Η ερώτηση μου είναι η εξή. Ε, στη Βαρσοβία παρατηρήσετε κάποια ένδειξη, κάποιο ότι θα ληφθεί κάποια απόφαση βάσει κάποιων σημείων αναφορά κάποιων κριτηρίων. Ή είμαστε έτοιμοι να δούμε ε, ελεύθερες δεσμεύσεις χωρίς σωστή βάση από τα κράτη-μέλη, γιατί χρειαζόμαστε αυτά τα σημεία αναφοράς. Χρειάζεται να λάβουμε υπόψη τις ε, διαφορετικές αυτές περιστάσεις στις διάφορες χώρες. Αυτό δεν συνέβη στη Βαρσόβια. Η Κίνα, η Ιαπωνία, ο Καναδάς ε, και οι άλλες χώρες ε, πρέπει και αυτές να συμμετέχουν στη συμφωνία και θα είναι δύσκολη η επιτεύξη αυτής της συμφωνίας στο Παρίσι. Εάν στο Παρίσι η Κίνα πει ότι θα μειώσει τις εκπομπές της κατά 10% εσείς θα μείνετε ικανοποιημένος ή θυμωμένος ή έκπληκτος οι συγκλονισμένε, Ποια θα είναι η αντίδρασή σα. Θα υπάρξουν πολλέ δεσμεύσει, πολλέ συμφωνίε. Εγώ έρχομαι από την Πολωνία και θέλω να κάνω έκκληση προ σας, να διαμαρτυρηθώ, να πω ε, μεγαλόφωνα ότι δεν πρέπει να μιλάμε αρνητικά για τα επιτεύγματά μα γιατί πολλά επιτύχαμε, έχουμε επενδύσει πολλά στην Ευρώπη. Επενδύουμε και στο κάρβουνο, αλλά αυτό το κάρβουνο είναι διαφορετικό. Η ενέργεια είναι πολύ ακριβή. Θα ήθελα να το πω στους σοσιαλιστές πρέπει να λάβετε υπόψη και το κοινωνικό, ε, την κοινωνική διάσταση. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τις κοινωνικές συνθήκες. Ξέρω ότι οι στόχοι μας είναι φιλόδοξοι, αλλά και τα κοινωνικά ζητήματα είναι πολύ σημαντικά και πολύ συχνά τα νοικοκυριά ξοδεύουν το 40% του οδήματός τους ε, για την ενέργεια. Αυτή είναι η κατάσταση η οποία επιδεινώνει τα ε, προβλήματα. Έχει προφανώς νόημα να ε, εξετάσουμε την κατάσταση δεδομένου ότι συνεχίζουν οι εισαγωγές ορυκτών καυσίμων προς την Ευρώπη. Πρέπει λοιπόν να δούμε όχι τι μας χωρίζει αλλά τι μας ενώνει. Υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη τα οποία αναφέρονται σε διαφορές μόνο, εγώ νομίζω ότι πρέπει να κοιτάξουμε πιο πολύ όχι τους διαχωριστικούς φραγμούς, αλλά τα σημεία συνάντησης, τα σημεία όπου συμφωνούμε. Ε, εκεί πρέπει να δώσουμε την έμφαση. Νομίζω ότι είχα κλείσει τον κατάλογο, αλλά αν ο κύριο Σόνικ θέλει ή να λάβει το λόγο, ε, ήρθατε μόλι τώρα νομίζω, ίσω δεν έχετε ακούσει κιόλα τι είπε ο Υπουργό, αλλά παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω μία ερώτηση. Θα ήθελα να απευθύνω στον Υπουργό. Κατηγορείται η Πολωνία ως ε, επενδύει υπερβολικά στον άνθρακα, ενώ επιβραδύνεται η παραγωγή στην Ευρώπη γενικότερα αληθεύει ότι η Γερμανία καίει τρεις φορές περισσότερο ακάρβουνα από ότι η Πολωνία. Αληθεύει ότι οι εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα στη Γερμανία αυξάνονται κατά τη διαστολή με αυτό που συμβαίνουν στην Πολωνία. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει ότι υπεγράφει η συμφωνία, η σύμβαση συνανασπισμού έχουμε υπογράψει ένα 60% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και θα ήθελα επίσης να πω ότι θετικό βρίσκω το ότι έγινε συζήτηση και στην Πολωνική Γερουσία. Ήμασταν παρόντε μαζί με συναδέλφου, εμεί η αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου. Ο κύριο Σιμάνσκι μιλήσαμε νομίζω με ειλικρίνεια. Συνομιλήσαμε με ειλικρίνεια. Ήταν πολύ καλή συνάντηση για όλου. Νομίζω ότι θα πρέπει να συζητάμε συχνά για τα θέματα αυτά και επίσης εγώ ως Γερμανός αλλά όλοι πρέπει να γνωρίζουμε γιατί έχει πολύ μεγάλη την πρώτη προτεραιότητα για την Πολωνία η ασφάλεια στην προμήθεια σε ενέργεια και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε όλη αυτή την ανταλλαγή απόψεων, σε όλο αυτό το διάλογο, το να απευθύνουμε κατηγορίες ο ένας τον άλλον δεν είναι καθόλου ευφιές. μόνο να δυναμητήσει την ατμόσφαιρα και τη συζήτηση μπορεί και πάντως δεν βοηθάει κανέναν. Και ξέρω ότι σαν συμπρόεδρος δεν είναι, ως, συμπρόεδρος δεν μπορεί να έχει κανείς τέτοιο έργο, να έχει ευχερές έργο όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Όπως είπα, η εξαποστάσεως θέρμανση στην Πολωνία έχει πολύ πολύ προχωρήσει, έχει υποδειγματική ανάπτυξη και αυτά τα θετικά σημεία θα πρέπει νομίζω να τονίζουμε και όχι αυτά στα οποία διαφωνούμε. Έχετε το λόγο παρακαλώ κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στις ερωτήσεις με τη σειρά με την οποία υπευλήθησαν. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω. Χθες επίσημα η πολεμική κυβέρνηση άλλαξε. αν Σχηματίστηκε Οπότε ο κ. ο Υπουργός Περιβάλλοντος ε, στο νέα σύνθεση υπουργών. Δημιουργήθηκε μια νέα λειτουργία, μια νέα θέση. Η θέση του υπευθύνου της πολιτικής κυβέρνησης, του πλερεξούσιου της πολιτικής κυβέρνησης για κλιματικά θέματα και αυτό το άτομο θα ασχολείται με τις διάφορες δραστηριότητες σε αυτό το τομέα. Και ο Πρωθυπουργός υπέγραψε το διορισμό μου ως Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Θα είμαι Γενικός Γραμματέας λοιπόν και πλήρε για την κλιματική πολιτική στην πολωνική κυβέρνηση. Αυτή είναι η βέλτιστη λύση κατά την άποψή μου. Η καλύτερη δυνατή για ποιο λόγο, διότι ένας άνθρωπος αρμόδιος για αυτή τη διαδικασία σε παγκόσμιο επίπεδο έχει πολλές δραστηριότητες πρέπει να έχει επαφές με τη γραμματεία της ε, συνθήκης, να βρίσκεται συναντήσεις που οργανώνονται στο πλαίσιο αυτών των παγκοσμίων διασκέψεων και πιθανώς θα γνωρίζετε ότι η εσωτερική κλιματική πολιτική παίρνει επίσης πάρα πολύ χρόνο, διότι στην Πολωνία έχουμε τη μεταρρύθμιση της νομοθεσίας περί υδάτων, τη μεταρρύθμιση της διαχείρισης αποβλήτων στην Πολωνία και φέτος στην Πολωνία επίσης προετοιμάζουμε μια νομοθεσία για το σχιστολιθικό φυσικό αέριο. Ο νέος Υπουργός, κ. Γκραμπόσκι, θα ασχοληθεί με αυτά τα εγχώρια ζητήματα. Και ξεχωριστά από αυτόν δημιουργείται μια θέση πληρεξούσου για το κλίμα. Και έτσι θα μπορώ εγώ να αφιερωθώ 100% στις ευρωπαϊκές συζητήσεις και στις παγκόσμιες επαφές και συζητήσεις σε επίπεδο συνθήκης η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω να σας ευχαριστήσω για θετικά σας σχόλια όσον αφορά τη διάσκεψη στη Βαρσοβία. Θα ήθελα να πω ότι λίγο καιρό πριν τη διάσκεψη η Πολωνία αξιολογήθηκε και θεωρήθηκε ότι πρόκειται για τη χώρα που καθυστερεί την Ευρώπη, ότι προσπαθεί να πνίξει την όλη διαδικασία το ότι οριστικοποιήσαμε τη διάσκεψη 24 ώρες αργότερα από ό,τι είχε προβλεφθεί μετά από πολλές ε, διαπραγματεύσεις και μια ε, νύχτα χωρίς να κοιμηθούμε. Πιστεύω ότι αυτό αποδεικνύει το ότι είμαστε αποφασισμένοι. Και στην Πολωνία είμαστε αποφασισμένοι να συμμετέχουμε σε αυτή την παγκόσμια διαδικασία. Θέλουμε να οριστικοποιηθούν όλα, να ολοκληρωθεί επιτυχώς αυτή η διαδικασία στο Παρίσι. Θέλουμε η συμφωνία στο Παρίσι να έχει μια νέα αξία. Θα θέλαμε αυτή η διασκέψη στο Παρίσι να εφαρμοστεί, να υλοποιηθεί και στις 194 χώρες. Θα θέλαμε να διαπραγματευτούμε μια συμφωνία στο Παρίσι η οποία θα επικυρωθεί επίσης και από 194 χώρες γιατί θέλω να σας υπενθυμίσω εκείνη την άσχημη εμπειρία που είχαμε στην πρώτη περίοδο του Κιώτο και την ακόμη χειρότερη εμπειρία όσον αφορά τη δεύτερη περίοδο του Κιώτο. Η δεύτερη περίοδος ε, περιορίζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Αυστραλία και μερικές χώρες του ΕΟΧ. 40% δηλαδή των παγκόσμιων ε, εκπομπών και η πρόκληση που έχουμε μπροστά μας είναι να αντιμετωπίσουμε το 100% των παγκόσμιων εκπομπών και μία, ένα από τα επιτεύγματα της συνάντησης ε, στη Βαρσόβια είναι ότι έχουμε έναν οδικό χάρτη και στη Λίμα θα έχουμε τα πρώτα σχέδια συμφωνίας. Στη Λίμα επίσης θα ορίσουμε τη μέθοδο υποβολής των συμβολών μας μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2015. Θα υποβάλουμε λοιπόν αυτές τις συμβολές μας το 2015 το πρώτο τρίμηνο ώστε να έχουμε πάρει χρόνο να προλάβουμε να ετοιμάσουμε τη συμφωνία ώστε το Παρίσι να είναι επιτυχές. Όσον αφορά την ευρωπαϊκή ατζέντα, ναι, πιστεύω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε ε, να μελετάμε το ποια θα είναι η ευρωπαϊκή συμβολή. Τι μορφή θα έχει. Πρέπει να σκεφτούμε τι επίπεδο φιλοδοξίας θέλουμε, πώς θα επιδιώξουμε να επιτύχουμε τις φιλοδοξίες αυτές ποια θα είναι η συμβουλή των επιμέρους κρατών μελών στη συνολική συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ποιο θα είναι το μεριδιό τους. Όλα αυτά τα ερωτήματα είναι πολύ σημαντικά και θα πρέπει να ξεκινήσουμε τώρα την περίοδο προβληματισμού μας. Ευτυχώς ε, έχουμε ένα χρόνο μπροστά μας, διότι τις συμβουλές μας θα πρέπει να τις παρουσιάσουμε στο πρώτο τρίμηνο του 2015. Ρωτήσατε επίσης για τις φιλοδοξίες μέχρι το 2020. Πολύ καλή ερώτηση, αιτιολογημένη και κατανοητή, διότι όσο περισσότερα κάνουμε μαζί ως διεθνής κοινότητα πριν το 2020, τόσο ευκολότερο θα είναι να υλοποιήσουμε τις πολιτικές μας μετά το 2020. Και αυτή η συζήτηση για το επίπεδο συμβολής ε, πριν το 2020 είναι πολύ σημαντική. Είναι πολύ σημαντική γιατί η δεύτερη περίοδος του Κιώτο περιορίστηκε σε κάποιες τρίτες χώρες και περίπου 160 χώρες βρίσκονται εκτός του συστήματος. Ε, πιστεύω λοιπόν ότι η ερώτηση σας είναι ε, πολύ σωστή εμείς ως διεθνής κοινότητα έχουμε φιλοδοξία σε αυτό το τομέα ή όχι. Και συμφωνώ μαζί σας ότι πρόκειται για μια πολύ σημαντική ερώτηση. Θα λάβει χώρα μια ξεχωριστή συνάντηση για το θέμα αυτό στη Βόνη στα μέσα του έτους όπου θα προσπαθήσουμε να βρούμε μια απάντηση σε αυτό το ερώτημα στη Βόνη. Θα ήθελα τώρα να αναφερθώ στα όσα είπε Θέλω να διαφωνήσω με ένα από τα πράγματα που είπατε. Είπατε ότι άλλαξε η γλώσσα και άλλαξε η συμβολή και αυτό αποτελεί οπισθοχώρηση. Εγώ διαφωνώ μαζί σας. Η απόφαση της Βαρσοβίας είναι 100% συμβατή με την απόφαση στον Τέρμπαν. Η απόφαση του Τέρμπαν λέει Η απόφαση του Ντέρμπαν ε, λέει ότι το 2015 η συμφωνία θα πρέπει να λάβει μια νέα διάσταση. Η συμφωνία αυτή θα περιλαμβάνει όλες τις χώρες και η λέξη contribution, συμβολή, αναφέρεται τόσο στις αναπτυσσόμενες όσο και στις αναπτυγμένες χώρες. Υπό αυτή την έννοια είναι 100% συμβατή με την αποφάση του Ντέρμπαν. Εάν επιλέγαμε άλλη διατύπωση, ανάλογα με την ομάδα χωρών για την οποία μιλάμε, αυτό θα σημαίνει διαφορετικό επίπεδο δεσμεύσεων και δεν θα υπήρχε έτσι, συνοχή με το πνεύμα της αποφάσης του Ντέρμπαν. Διότι πρέπει να διαπραγματευτούμε, καλούμαστε να διαπραγματευτούμε μια συμφωνία η οποία θα ισχύει για όλους αυτός ο όρος λοιπόν contribution, συμβολή, είναι πολύ σημαντικός, εξυπηρετεί το σκοπό που θέλουμε και είναι ένα από τα επιτεύγματα της Βαρσοβίας διότι η συμφωνία που εμείς διαπραγματευόμαστε πρέπει να προσκαλεί τους ανθρώπους όχι να είναι αποτρεπτική συμφωνία, να μην θέλουμε χωρίς να συμμετάσχουν σε αυτό. Αυτές οι συμβολές φυσικά μπορούν να έχουν διάφορες μορφές, μπορεί να είναι πολιτική, δασική, μπορεί να είναι πολιτική ενεργειακή απόδοση ή ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κάποιο είδους φόρος ε, διοξιδίου του άνθρακα στα σύνορα για παράδειγμα συνεπώς η φύση της συμβολής της ε, εκάστοτε χώρας ε, θα είναι διαφορετική δεν θα έχουμε την ίδια συμβολή για τον καθένα, για το κάθε μέρος, διότι κάποιες χώρες είναι διπλάσιες σε μέγεθος από την Ευρώπη και υπάρχουν άλλες χώρες που είναι μικρότερες από τις Βρυξέλλες. Δεν μπορούμε λοιπόν να έχουμε μία, ε, την ίδια επιλογή, την ίδια λύση για όλους. Θα πρέπει να έχουμε ένα τεράστιο εύρος λύσεων που να μπορεί να εφαρμοστεί στα διάφορα κράτη. Όσον αφορά τώρα το 30% έχουμε λάβει μια πολιτική απόφαση στην Ευρώπη για το 30%. Το 30% είναι αυτό που προσφέρουμε. Αυτό βάζουμε στο τραπέζι. Αν επιτευχθεί η παγκόσμια συμφωνία και οι υπόλοιπε οι επωνομαζόμενες ανεπτυγμένες χώρες ε, κάνουν παρόμοιες προσπάθειες αυτή η απόφαση λήφθηκε το 2007 και όλα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρονται σε αυτή την ε, απόφαση του 2007. Πιστεύω δεν υπάρχει λόγος λοιπόν να το επαναλαμβάνουμε ξανά και ξανά. Όσον αφορά τις συμβολές, ε, τη χρηματοδότηση για το Ταμείο Προσαρμογής ε, καταφέραμε να συλλέξουμε 100 εκατομμύρια και όχι 80 θα ήθελα να πω ότι εγώ έχω εντυπωσιαστεί από κάποιες μονομερείς δεσμεύσεις ε, χρηματοδότησης. Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Νορβηγία, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η ΕΠΑ, η Κορέα, η Ιαπωνία, η Σουηδία, η Γερμανία, η Φιλανδία και οι κατοχώρες. Με έχει εντυπωσιάσει η προσφορά που έκαναν. Και ήταν εθελοντική αυτή η προσφορά. τεράστια συμβολή σε αυτή την οικονομική πτυχή της κλιματικής ε, πολιτικής. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Γκέρα για την ερώτησή του. Θα ήθελα να πω ότι το σημαντικότερο μας καθήκον στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων της Συμφωνίας του Παρισιού θα είναι να αποφύγουμε αυτήν, αυτόν τον κίνδυνο ενός τρίτου Κιώτο, διότι η λογική του Κιώτο ήταν ότι έχουμε δύο χωριστά διαμερίσματα. Από τη μια έχουμε τις ανεπτυγμένες χώρες και από την άλλη τις αναπτυσσόμενες. Αλλά εμείς εδώ δεν μπορούμε να προσπαθούμε να χτυπήσουμε το 14% των εκπομπών, αλλά το 100%. Το σημαντικότερο θέμα τώρα εδώ είναι πώς θα δημιουργηθεί, τι μορφή θα έχει ένα τέτοιο μηχανισμό, πώς μπορεί να δημιουργηθεί αυτή η μέθοδος η οποία θα είναι ανοιχτή σε όλα τα μέρη. Μελετώντα τη συνθήκη, η συνθήκη αυτή δημιουργήθηκε από το αποκύμα του ε, διάσκεψης για τη ιστορία, για τη βιώσιμη ανάπτυξη και στόχος της συνθήκης ήταν ε, η μείωση των εκπομπών, η εξάλληψη των εκπομπών, αλλά ταυτόχρονα η συνθήκη παροτρύνει για βιώσιμη ανάπτυξη και καταπολέμηση της φτώχειας. Αυτή είναι η κύριη στόχη της συνθήκης. Εμείς θα πρέπει να εκπονήσουμε τη συμφωνία με τέτοιο τρόπο να είναι διατυπωμένη συμφωνία με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί από την Ευρώπη, από το Κυριμπάτι, από τα νησιά Κυριμπάτι, από τι Ηνωμένε Πολιτείε, από τη Ρωσική Ομοσπονδία και από την Κίνα, από την Τουβαλού και από την Ινδία και από ένα σωρό άλλε χώρε. Είναι πολύ δύσκολο καθήκον, πολύ δύσκολο έργο, αλλά πιστεύω ότι με αμοιβαία εμπιστοσύνη εφόσον δείξουμε εμπιστοσύνη οι μεν στους δε, είναι δυνατή η συμφωνία. Επίσης τέθηκε το ερώτημα του ρόλου των μη κυβερνητικών οργανώσεων στη Βαρσοβία. Οι ενώσει, οργανισμοί, μη κυβερνητικοί που ασχολούνται με το κλίμα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία γιατί κοινοτοποιούν την κοινή γνώμη παρέχουν κίνητρα στις κυβερνήσεις να επιτείνουν τις προσπάθειές τους όσον αφορά την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Να σας υπενθυμίσω ότι ορισμένες από αυτές με κυβερνητικές οργανώσεις δύο-τρεις από αυτές δήλωσαν ότι η διάσκεψη της Βαρσοβίας θα να φιάσκω 24 ώρες πριν καν κλείσει, πριν ολοκληρωθεί. Και σας πενθυμίζω ότι τελείωσε η διάσκεψη με 24 ώρες καθυστέρηση σε σχέση με το ότι είχε προβλεφθεί. Συνεπώς ε, κάποιοι τέτοιοι μη κυβερνητικοί οργανισμοί είχαν εγκαταλείψει τους χώρους της διάσκεψης 24 ώρες, 48 ώρες ουσιαστικά πριν ε, Ισχυριζόμενος ότι δεν έβλεπαν κανένα αποτέλεσμα, δεν επιτεύχθηκαν κανένα αποτέλεσμα. Νομίζω ότι είναι αυταπόδεκτο το υπόλοιπο. Ε, δεν, δεν υπάρχει λόγο να το συζητήσουμε περαιτέρω. Ε, κύριος Τσαμάσκιν, ερώτησή σας. Ε, θα ήθελα να σε επιβεβαιώσω. Όσα είπα κατά την παρουσίασή μου εδώ στην Επιτροπή αυτή. Ναι, πρώτα απ' όλα έχουμε μια παγκόσμια συμφωνία. τέτοιου είδους συμφωνία θέλουμε να υπογράψουν και να επικυρώσουν και οι άλλες ανεπτυγμένες χώρες, όχι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ανεπτυσσόμενες χώρες, θέλουμε να συμμετάσχουν και οι λοιπές ανεπτυγμένες χώρες. Αυτή η ενεργειακή πολιτική που βλέπουμε πέραν της Ευρώπης ε, στην Αμερική με ενέργεια χαμηλής χαμηλού κόστους και μείωση εκπομπών ταυτόχρονα θα έπρεπε να μας εμπνεύσει στις συζητήσεις που κάνουμε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επανάσταση του σχιστολίθου στις Ηνωμένες Πολιτείες ε, καθιστά τις Ηνωμένες Πολιτείες ε, απολύτως αυτόνομες ε, δεν εξαρτώνται πλέον τόσο πολύ από τι εισαγωγέ ορυκτών καυσίμων, γιατί αυτό είπατε κύριε Πρόεδρε, πρέπει να είμαστε ανεξάρτητοι και οι Αμερικανοί χάρη στην επανάσταση του σχιστολιθικού αερίου και πετρελαίου κατάφεραν να είναι ανεξάρτητοι, αλλά κατάφεραν και άλλα δύο πράγματα. Μείωσαν την τιμή τη ενέργεια και επίση μείωσαν και τι εκπομπέ. οι οποίε ήταν οι ήταν διπλάσια η μείωση από τις φιλοδοξίες της δικές μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν μιλήσαμε στους εκπροσώπους του τομέα και μιλάμε και για επενδύσεις σε τομείς ε, υψηλής κατανάλωσης ενέργειας, ε, λένε ότι ε, τα δολάρια που θέλουν να επενδύσουν θα τα επενδύσουν αλλού και όχι εδώ στην Ευρώπη ή στη μιση Ανατολή ή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πιστεύω ότι τη σημερινή μέρα όταν μιλάμε για παγκόσμια κρίση γνωρίζουμε ότι δεν είναι παγκόσμια, είναι ευρωπαϊκή. Αυτά τα σχόλια ε, της βιομηχανίας θα πρέπει να ληφθούν πολύ στα σοβαρά. Θα ήθελα επίσης να απαντήσω στα όσα είπε ο Δεν έχω λεπτομερή στοιχεία για τους επιμέρους, ε, τα επιμέρους επίπεδα εκπομπών των κρατών μελών. Θα μπορούσατε να κάνετε αυτή την ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παράσχει στατιστικά στοιχεία για τις εκπομπές των ε, κρατών μελών και να μας πει πού παρατηρείται το χαμηλότερο ποσοστό εκπομπών, πού αυξάνονται οι εκπομπές. Ε. και σε σχέση με το ΑΕΠ των χωρών αυτών. Και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να εικονίσει τέτοιε στατιστικέ. Νομίζω ότι τέτοια στατιστικά στοιχεία για τα επόμενα δύο-τρία χρόνια θα μπορούσαν να μας ωφελήσουν ιδιαίτερα στις εσωτερικέ μα συζητήσει. Δεν γνωρίζω όμω τα πάντα για το θέμα αυτό και δεν θέλω να δημιουργήσω κάποιο σύγχυση Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως ανεξάρτητος φορέας θα μπορούσε να παράγει τέτοια στοιχεία για τα τελευταία δύο-τρία χρόνια. Ναι, πράγματι, οι πληροφορίες αυτές θα παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Αλλά δεν θα ήθελα αυτή τη στιγμή να σχολιά, τη σχολιάσω, γιατί πιστεύω ότι για να σχολιάσουμε πρέπει να βαζόμαστε σε αξιόπιστα και ρεαλιστικά δεδομένα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση λιθάρθρακας, τέραβατ, αναώρα, μέχρι το 2012 με τον λιθάρθρακα έχουμε 17 τέραβατ ε, την ώρα, ανα, ε, τεραβατόρα για την πρώτη περίοδο. Εν πάση περιπτώσει έχουν, έχει γίνει αντιστάθμιση, αλλά θα μας δώσει τις λεπτομέρειες η Επιτροπή φαντάζομαι. Η Επιτροπή παρακαλώ. Ευχαριστώ και ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να επανέλθω σε αυτό το ζήτημα. Αν δείτε τελευταίες, ε, τα τελευταία στοιχεία για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που δημοσιεύθηκε πριν από λίγο από την Ευρωπαϊκή Περιβαλλοντική Υπηρεσία, σελίδα 10 της έκθεσης ε, και την, την ε, σύνοψη θα δείτε τα profiles για όλα τα μεμονωμένα κράτη-μέλη. Ας δώσω ένα παράδειγμα, η αλλαγή σε εκπομπές στη Γερμανία από το 2010 μέχρι το 2011 υπήρξε μείωση 2,9%. Να σας πω και σε άλλα κράτη-μέλη Υπάρχουν πολλά παραδείγματα, αλλά μπορείτε να τα βρείτε σε αυτή την έκθεση και στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Περιβαλλοντικής Υπηρεσίας. Ευχαριστώ πολύ. Έτσι κλείνει η συζήτηση. Έχουμε κάποια θέματα να συζητήσουμε ασφαλώ. Η ατμόσφαιρα των συστήσεων ήταν καλή. Έχουμε να σημειώσουμε και κλιματική αλλαγή εδώ και πιστεύω ότι θα καταφέρουμε για τα 500 εκατομμύρια των Ευρωπαίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εξασφαλίσουμε ένα μέλλον ασφαλές οικονομικά, οικολογικά, κοινωνικά. Αυτό προσπαθούμε όλοι. Αυτό επιδιώκουμε. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία κύριε Κορόλετς για τις επόμενες ημέρες, εβδομάδες, μήνες στη νέα δουλειά σας, στην τριμερή αυτή προεδρία και φαντάζομαι στο Παρίσι θα έχουμε εν τέλει να σημειώσουμε μια νίκη που χρειάζεται τόσο πολύ ο κόσμος γιατί έχουμε το στόχο του 3,7 να επιτύχουμε εμείς η παγκόσμια κοινότητα προτίμησε το 2 ως στόχο πώ χρειάζονται περισσότερες προσπάθειες, αλλά γι' αυτό είμαστε εδώ, γι' αυτό και συνεργαζόμαστε και εύχομαι κάθε επιτυχία. Όπως είπα, ευχαριστώ και πάλι που ήρθατε και ξέρω ότι θα έχετε πολύ και σκληρή δουλειά για τι επόμενε για τις επόμενες εβδομάδες και μήνες. Jetzt Και τώρα συνεχίζουμε. Στο επόμενο θέμα της ημερησίας διατάξεως. Και έχω την πολύ μεγάλη χαρά να συζητώ... Α, να έχω τον κύριο Σανώνη. Με τον ένα συνάδελφο και τις κυρίες συναδέλφους. Έχουμε μόνο κυρίε εκτός από τον κύριο Τσανώνη. Για την ανταλλαγή αυτή με την Επιτροπή και την ΕΑΤ σχετικά με τα γενετικά τροποποιημένα ζώα. Καλώς ήρθατε τον κύριο Κολέ τη Επιτροπή. Του δίνω πρώτα το λόγο και μετά από την ΕΑΤ, η κυρία Βίτμαν. Παρακαλώ. Κύριε Πούλε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Η συζήτηση που έχουμε σήμερα είναι μια σοβαρή συζήτηση, ενδιαφέρουσα συζήτηση, σημαντική και ως προς τις πολιτικές αλλά και ως προς τις περιβαλλοντικές της διαστάσεις. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε μάλλον τη συζήτηση, την συνήθεια να υποβάλουμε προς έγκριση φυτά. Το πρόβλημα των ζώων είναι σχετικά καινούριο, εκτός από ένα σημείο, στο οποίο θα αναφερθώ βέβαια, αλλά ξέρετε ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε εδώ και χρόνια έχουν αναπτύξει σολομό γενετικά τροποποιημένο ο οποίος με τα γονίδια που του έχουν μεταβιβαστεί στο γενετικό του υλικό ε, διπλασιάζει το βάρος του, ε, μάλλον αυξάνει το βάρος του με ρυθμούς διπλάσιους από τον κανονικό σολομό και η FAO, η Food and Drug Administration στις ΗΠΑ αξιολογεί τους κινδύνους για την ανθρώπινη, για τη δημόσια υγεία από τη διατροφή με τέτοιου είδους ε, σολομούς. Η FDA λοιπόν δίνει μια σειρά από γνωμοδοτήσεις για τον γενετικά τροποποιημένο αυτό οργανισμό, ε, τον Σολομό, ο οποίος ακόμη δεν έχει τεθεί στην αγορά των ΗΠΑ. Η ανάπτυξη του έγινε παράλληλα και στον Καναδά, σε ηχθείο τροφία, ε, σε μορφή γόνου καλύτερα στον Καναδά και στις ΗΠΑ σε τροφία. Είναι κάτι που μας αφορά ασφαλώς, διότι ε, εξάγουν από, ε, προς εμάς οι Ηνωμένες Πολιτείες Σολομό. Βέβαια πρόκειται για Σολομό ελεύθερης βοσκής από το Ιναλάσκα κυρίως σε ε, κονσέρβα και πολύ πιο σπάνια για Σολομό εχθειοτροφίου. Ο Σολομός εχθειοτροφίου είτε από την Νορβηγία είτε από τη Χιλή προέρχεται και μπαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά θέλησαμε να προλάβουμε το ενδεχόμενο να υποβληθεί επίσημο αίτημα για τη διάθεση του κρέατος αυτού του γενετικά τροπημένου ε, σολομού στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή για την είσοδο ζών των ζών, ζών των σολομών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι λοιπόν, ούτε για σάρκα, ούτε για ζώντες σολομούς έχουν υποβληθεί ακόμη αιτήσει, αλλά εμείς θελήσαμε να προλάβουμε και ζητούμε από την ΕΑΤ, την ΕΣΑ την επιστημονική μας ε, υπηρεσία να ε, ετοιμάσει τις απαιτήσεις, τις επιστημονικές ώστε να είμαστε έτοιμοι σε περίπτωση που ζητηθεί η ευρωπαϊκή άδεια να είναι το τεχνικό δελτίο, ο φάκελος με τις προϋποθέσεις μας και τις απαιτήσεις έτοιμες, έτοιμος για όποια ε, επιχείρηση ενδεχομένω θέλει να εισαγάγει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ έχω την εκπρόσωπο τη ΕΑΤ, η οποία μπορεί να σα δώσει τι εξηγήσει, εάν θέλετε, για τι απαιτήσει που έχουν ε, οριστεί. Έχουμε επίση τον εκπρόσωπο τη Γενική Διευθύνσεω Έρευνα. Α, δεν τον βλέπω που πήγε. Α, εκεί πίσω πήγε, συγγνώμη. Ε, υπεύθυνο του προγράμματο Πίγασο, Πέγκαζιου. Και ο οποίο, αν θέλετε, θα σα δώσει εξηγήσει για το πρόγραμμα. Αν μου επιτρέπετε όμως κύριε Πρόεδρε, θα παρακαλούσα να επιτραπεί στην ΕΦΣΑ, στην ΕΑΤ, να δώσει εξηγήσει για τις προϋποθέσεις στο θέμα του Σολομού. Ευχαριστώ κύριε Πούλε, λέει ο Πρόεδρος, πολύ ευχαριστώ. Καταρχάς ευχαριστώ για τις παρουσιάσεις εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, πολύ φρόνιμη αυτή η, η πρόσκληση να δώσουμε το λόγο στην ΕΑΤ. Παρακαλώ κύριε Βάιτμαν. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομη δεν έχουμε πολύ χρόνο. Η ΑΤ έχει εκδώσει δύο έγγραφα κατευθύνσεων για τις πτυχές ε, τροφίμων και ασφάλες... όπως και δημόσιας υγείας και ένα για την αξιολόγηση περιβαλλοντικών κινδύνων σε περίπτωση που ε, προκύψει απελευθέρωση ζώντος ζώου στο ευρωπαϊκό περιβάλλον. Οι κατευθύνες γραμμές αυτές ακολουθούν τις ίδιες αυτές αρχές που έχουμε για την αξιολόγηση των γενετικά τροπημένων φυτών. Επικεντρωνόμαστε λοιπόν σε μια συγκριτική προσέγγιση. Συγκρίνουμε το γενετικό τροποποιημένο ζώο σε ένα ισοδύναμο μη γενετικό τροποποιημένο ζώο του ίδιου είδους και προχωρούμε βέβαια στα βήματα όπως ακριβώς και με τα ε, φυτά, τα γενετικά τροποποιημένα, δηλαδή κοιτάμε τα μοριακά χαρακτηριστικά, την αξιολόγηση του κινδύνου, τη συγκριτική προσέγγιση που είναι το επίκεντρο αυτής της αξιολόγησης κινδύνου, δηλαδή το καθεστώς υγείας, ευημερίας, κοινωνικής συμπεριφοράς, σύνθεση των διαφόρων ιστών, οργάνων, προϊόντων του εν λόγω ζώου, αν ο λόγος βεβαίως και της τροποποίησης, και, την, και η έκβαση αυτού του συλλογικού ε, πακέτου αξιολόγηση και δεδομένων θα προχωρήσει σε μια αξιολόγηση για το τι είδους μελέτες αλλεργιολογικές, διατροφικές και το καθεξής ενδεχομένως χρειαστούν. Και... Μια και έχουμε ασχοληθεί με το θέμα της υγείας του ζώου και της ευημερίας του, θα ήθελα να δώσω πιο πολλές λεπτομέρειες σε αυτό. Στην φάση της ανάπτυξης, ήδη δηλαδή στο εργαστήριο αυτό του γενετικά τροποποιημένου ζώου, πριν από τη γέννηση ξεκινάει η αξιολόγηση της υγείας του και της ευημερία του και μέσα στο εργαστήριο μετά τη γέννηση και στο περιβάλλον το ελεγχόμενο της εκμετάλλευσης με, άλλο, με άλλα ζώα του ιδίου ίδιου, είδους, με την κοινωνική συμπεριφορά δηλαδή του ζώου που παρακολουθείται στενά και μετά έχουμε μια θα λέγαμε δοκιμή κλινική ούτως υπήν, δηλαδή παρακολουθούμε ε, τις παραμέτρους αυτές της υγείας και της ευημερίας και τις φυσιολογικές παραμέτρους και τη συμπεριφορά του ζώου με δεδομένα τα οποία εισάγονται μετά στο κεντρικό πακέτο δεδομένων ώστε αν έρθει ποτέ μια τέτοια αίτηση στην ΕΑΤ να έχουμε τις απαιτήσει μας έτοιμες. Αυτά έχω να πω προς το παρόν, αν τυχόν υπάρχουν από τις ερωτήσεις, πολύ ευχαριστώ να διευκρινίσω. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Η έτερη Γενική Διεύθυνση, παρακαλώ, έρευνα. Να μας κάνετε την παρουσίαση. Η παρουσίαση είναι διαθέσιμη, επαναλαμβάνω, και στην, ε, στο, στο, τοπό μας. Ε, έχουμε και το web streaming για όποιον θέλει να παρακολουθήσει φυσικά θα υπάρχει δυνατότητα. Ευχαριστώ που μου επιτρέπετε να παρουσιάσω το πρόγραμμα Πήγασος ε, και τα βασικά πορίσματά του. Ε, υπάρχουν ε, λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα όπως είπατε και θα μπορούσα να σας δώσω και εδώ λεπτομέρειες αλλά επειδή δεν έχουμε χρόνο θα σας κάνω τη σύνοψη. Είναι ένα μικρό πρόγραμμα το Πήγασος που υποστηρίχθηκε χρηματοδοτικά από το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα για μία διετία, Αύγουστος 2009 έως Ιούλιος 2011. Έχει κλείσει, έχει περατωθεί το πρόγραμμα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ε, πρόκειται για μια συντονιστική δράση ουσιαστικά. Δεν υπήρξε έρευνα εργαστηριακή για γενετικά τροποποιημένα ζώα στα πλαίσια του προγράμματος. Εξετάζαμε ε, την κοινωνική η συμπεριφορά και τις οικονομικές επιπτώσεις ε, της ε, θέσης εμπορία των γενετικά τροποποιημένων ζώων. Στην ιστοσελίδα μπορείτε να δείτε συγκεκριμένα οικονομικά αποτελέσματα και όλες τις επιδόσεις ε, τα deliverables του προγράμματος δεν υπάρχουν όλα, υπάρχουν μόνο αυτά που συνιστούν δημόσιες πληροφορίες, τα υπόλοιπα μπορείτε κατόπιν αιτήματος να τα ε, λάβετε επίσης το πρόγραμμα εργασίας μας μετά από αίτημα της ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ασχολήθηκε με ένα ζήτημα ένα πολύ συγκεκριμένο ζήτημα. Ε, αυτό προέκυψε ε, και από μια κοινή σύσκεψη με τη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ ΣΑΝΚΟ. Οικονομικέ λοιπόν πτυχέ των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών για κάποιε πτυχέ τη πολιτική. Δεν εννοούμε καθόλου την νομοθεσία. Αυτό εντάσσεται μάλλον στην αξιολόγηση. Ε, ασχολούμαστε με ε, τα, την κοινωνική συμπεριφορά των ζών και θέματα που ε, απασχολούν περισσότερο ε, τους καταναλωτές. Έγιναν διάφορα εργαστήρια επίσης για να καλυφθούν οι ανησυχίες των εμπλεκομένων φορέων. Τρία εργαστήρια έγιναν κατά τη διάρκεια του προγράμματος στην Νορβηγία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία. Στις Βρυξέλλες έγινε ένα τέταρτο εργαστήρι όπου συμμετείχαν όλοι όσοι ενδιαφέρονταν για τη διάσταση της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης και τέλος στην Ινδία έγινε ένα εργαστήρι για να δούμε και την εξωτερική διάσταση εκτός Ένωσης Επίσης ε, ε, έγιναν ε, συζητήσεις πολιτών για να ακουστούν οι φωνές των εμπλεκομένων φορέων, τα citizen juries, τα λεγόμενα, το 2011 και 2012, ένα στο Ηνωμένο Βασίλειο και ένα άλλο στη Δανία. Για τα αποτελέσματα και τα βασικά πορίσματα και συστάσεις, θα έλεγα ότι ένα βασικό στοιχείο είναι ότι τα γενετικά τροποποιημένα ζώα θα πρέπει να εξεταστούν ε, κατά περίπτωση. Ε, οι αιτήσει που υποβάλλονται για τα γενετικά τροποποιημένα ζώα δεν δημιουργούν τα ίδια ζητήματα από ε, πλευρικής πλευράς, από ε, πλευράς διοντολογίας μάλλον ε, και ως προς τις άλλες πτυχές. Για τη μεθοδολογία και την αξιολόγηση των πιθανών επιπτώσεων Λαμβάνουμε υπόψη ταυτόχρονα και τις επιθυμίες ε, των πολιτών. Ε, ανιχνευσιμότητα και σήμανση είναι άλλα σημαντικά ζητήματα για τα τρόφιμα ε, σε όλες τις περιοχές όπου συλλέξαμε δεδομένα. Δηλαδή, έγινε με μια μετα-ανάλυση των δεδομένων περιοχή και από εκεί προκύπτουν αυτά τα συμπεράσματα. τα προθέματα, τα διοντολογικά για τους ε, καταναλωτές ε, ε, που μας θυμίζουν και ζητήματα που προκύπτουν και για άλλες ζητήματα βιοτεχνολογίας σχετίζονται με την ευημερία των ζώων και τις πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Αυτά είναι, αυτές είναι οι βασικότερες διοντολογικές ανησυχίες, το ότι μπαίνουμε στα χωράφια της φύσης και αλλάζουμε τη φυσική της πορεία. Όταν προσπαθούμε να θέσουμε σε πορεία και να χαράξουμε την πορεία ενός γενετικά τροποποιημένου ζώου. Όλα τα θεατολογικά ζητήματα πρέπει οπωσδήποτε να συνυπολογίζονται στην αξιολόγηση αντικτύπου, να συνεκτιμώνται. Οι σε εμπορία τροφίμων που προέρχονται από τέτοια ζώα. Ε, επίσης πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ανησυχίες των καταναλωτών κατά περίπτωση διότι ανάλογα με τις εφαρμογέ, τις εμπορικές εφαρμογές ε, ποικίλουν ε, και οι ανησυχίες. Ε, διότι μιλάμε μόνο για παραγωγή τροφίμων αλλά και βιοκαλλιέργειες το Είδα καλλιέργειε. Ε, εξατάστηκαν ε, τρία διαφορετικά σενάρια. Η θέση εμπορία πρέπει να λαμβάνει υπόψη το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο και την προσαρμογή του στην παγκόσμια διάσταση. Uh, ε, θα πρέπει επίσης να εκτιμήσουμε τις ε, πιθανές, ε, τα πιθανά ωφέλη και τους πιθανούς κινδύνους για, όταν μπαίνουν στην κυκλοφορία τα προϊόντα των γενετικά τροπημένων οργανισμών καθώς και τα ζητήματα όπως έλεγα τα διοντολογικά και οι οικονομικές επιπτώσεις της εμπορία σε αυτών των προϊόντων και σε ένα ορισμένο βαθμό θα πρέπει να υπάρχει μια επικοινωνία διαρκώ με τους καταναλωτές για την ισορροπία που πρέπει να επιτευχθεί ανάμεσα στα όφελη και τους κινδύνους ε, για την πιθανή είσοδο στην αγορά των προϊόντων των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, διότι δεν είναι πεπισμένοι απαραίτητα οι καταναλωτέ με την επιχειρηματολογία για την ισοδυναμία. Δηλαδή ότι τα νέα, τα novel foods, ε, τα νέα τρόφιμα είναι ισοδύναμα με τα παραδοσιακά. Αυτά είναι τα βασικά συμπεράσματα του προγράμματο. Ευχαριστώ για την παρουσίαση. Κύριε Μακέβον που έχετε τυπώσει την ερώτηση Λίντα, θέλεις να λάβεις εσύ πρώτη το λόγο ή τελευταία ενδεχομένω την προτιμάς. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα πρέπει δυστυχώς να αποχωρήσω στις 5. 5 παρα 20 για να προλάβω να γυρίσω στη Βόρεια Αγγλία σήμερα. Με όλα τα τρένα, τα αεροπλάνα, το στο ένα τρένο να πιάσω το άλλο τρένο κτλ. Ε, να προλάβω το άλλο τρένο. Ευχαριστώ λοιπόν τον ε, κύριο Πουλέ που έκανε την παρουσίαση. Ο Βρετανικός τύπος τη Δευτέρα λέει ότι ε, είπε ότι δόθηκε άδεια για εμπορική εκμετάλλευση γενετικά τροπημένων οργανισμών. Κάτι με τον Παναμά. Δηλαδή ότι δόθηκε σχετική έγκριση. Και μάλιστα λένε ότι η καναδική κυβέρνηση έδωσε μεν την άδεια λέγοντας ταυτόχρονα ότι για τα γενετικά τροποποιημένα ψάρια έχουν, να παρουσιάζουν μεγαλύτερο κίνδυνο διαφυγής στη φύση αλλά και ότι δεν προβλέπεται ε, άμεσα να διατεθεί στην αγορά για κατανάλωση το ψάρι αυτό. Δηλαδή δίνει μια άδεια για κάτι που θα γίνει στον Παναμά αλλά στο ιστορικό του ο Καναδάς λέει «Α, όχι, εμείς δεν το θέλουμε». Έχει αρχίσει πάντως ε, να παίζεται κάποιο παιχνίδι από ό,τι φαίνεται στην υπόθεση αυτή. Και καταλαβαίνω βέβαια ότι η έχει κάνει το καθήκον της. Με χαρά βλέπω ότι μιλούμε για ωφέλη και κινδύνους έτσι όπως τα προβλέπουμε ή τα διαβλέπουμε. Αλλά νομίζω ότι ξαναμπαίνουμε στη συζήτηση της κλωνοποίησης. Και το έχω ήδη πει στην Επιτροπή. Μιλούμε για ασφάλεια των τροφίμων, αν είναι ασφαλείς οι τροφές, αλλά εάν περιουστεί μόνο σε αυτό η ΕΑΤ, δεν θα ικανοποιήσει, δεν θα καθησυχάσει τους πολίτες, όσο απέτυχε και στην κλωνοποίηση θα αποτύχει και εδώ, γιατί γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί δεν αφορούν μόνο την ασφάλεια των τροφίμων. Εγώ δεν πιστεύω ότι αν φάω γενετικά τροποποιημένη τροφή θα πάθω κακό. Δεν υπάρχει τέτοιου είδους επιστημονική απόδειξη και δεν το πιστεύω. Αλλά δεν μας έχει πείσει κανείς ότι η χρήση γενετικά τροποποιημένων ε, οργανισμών, φερειπίνησης καλλιέργειας δεν μπορεί να επηρεάσει τη βιοπικιλότητα. Έχουμε δει στην Ινδία να επηρεάζεται από το ένα χωράφι στο άλλο η βιοπικιλότητα από μέρος στο οποίο καλλιεργούνται γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί σε άλλο που δεν επιτρεπόταν η χρήση τους. Αυτό είναι που απασχολεί τον πολίτη. Και στα πρόσθετα, στις πρόσθετες ουσίες, ερωτώ, την Επιτροπή και το έχω ξανακάνει. Τι έχει κερδίσει ο καταναλωτής σε σχέση με αυτό που είχε μέχρι τώρα. Τι κερδίζει παραδείγματι αν το συγκρίνουμε φερειπήρ στην ευημερία των ζώων. Έτσι. Δεν ξέρω αν αυτό έχει ήδη περάσει στην Επιτροπή Δεοντολογίας, γιατί το θέμα της κλωνοποίησης είχε πάει στην Επιτροπή Δεοντολογίας και έτσι δόθηκε η αρνητική απάντηση στις κλωνοποιημένες τροφές με το σκεπτικό ότι ήταν ε, πολλά τα ζητήματα δεοντολογίας που αφορούσαν το, την κλωνοποίηση και γι' αυτό δεν έπρεπε να μπει στην ε, διατροφική αλυσίδα. Το ίδιο πιστεύω θα πρέπει να γίνει και εδώ. Και βλέπω ότι δεν αντιλαμβάνεστε, δεν λαμβάνετε υπόψη την κοινή γνώμη στην υπόθεση αυτή. Γιατί είναι άλλο η αντίληψη που έχει κανείς για τη χρήση των γενετικά τροπημένων οργανισμών σε στροφές και άλλη στην ε, χρήση τους για έρευνα. Για μένα τουλάχιστον υπάρχει μεγάλη διαφορά γενετικά τροποποιημένα έμβρια. Όχι ανθρώπων, έτσι, ηχθείων, ηχθείων ε, γόνος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί, να καταστραφεί σε μερικές εβδομάδες μετά, που μας βοηθάει με την έρευνα αυτή να καταπολεμήσουμε ίσως τις πιο φρικτές αρρώσεις που ταλανίζουν το ανθρώπινο είδος, το δέχομαι αυτό εγώ. Άλλο είναι το να χρησιμοποιηθεί το ε, γενετικά τροποποιημένο αυτό έμβριο και άλλο το να, γι... εξετάσω την ευημερία του ζώου σε ένα ζώο που έχει γενετικά τροπηθεί και φερειπίν μου δίνει ένα γουρνάκι με πιο κοντά πόδια, με πιο μακρύ σώμα και δεν ξέρω τι. Άλλη υπόθεση αυτή. Και ευχαριστώ την Επιτροπή, αλλά πιστεύω ότι χρειάζεται ένα ευρύ και δημόσιο διάλογο. Δεν είναι ένα τεχνοκρατικό ζήτημα αυτό το οποίο μπορούμε να κλείσουμε με μια απλή συζήτηση εδώ στο Κοινοβούλιο ή σε ένα γραφείο κλειστό. Ούτως ή άλλως και στην επόμενη θητεία θα πρέπει να μας απασχολήσει αυτό. Ευχαριστώ κυρίο, ε, κυρία Μακέβαν. Η κυρία Πιλάρα Ιούσο που είναι και η συνάδελφος που έχει την επαφή, είναι πρόσωπο επαφής με την ΕΤΑ. Ακούμε την κυρία Λεπάζ, μετά τον κύριο Σλούτερ, την κυρία Κιόμ και το καθεξής. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την ΕΦΣΑ και την Κομισιόν που ήρθαν να μας μιλήσουν για το ζήτημα αυτό. Είναι ένα σημαντικό ζήτημα και πρέπει να ξεκινήσουμε τη συζήτηση τώρα. Αντιλαμβάνομαι πολύ καλά ότι η αποστολή της ΕΦΣΑ είναι να μας πει κατά πόσο αυτά τα γενετικώς τροποποιημένα ζώα μπορούν να καταναλωθούν με ασφάλεια και κατά πόσο συμμορφώνονται ή όχι με όλους τους κανόνες ασφάλειας των τροφίμων. Αλλά εδώ ουσιαστικά η συζήτηση είναι διτή. Όπως είχαμε με το κρέας, οι καταναλωτέ το θέλουν αυτό το κρέας ή όχι. Αυτή το, το ερώτημα ε, είναι δύο τελείως διαφορετικέ συζητήσει που πρέπει να επιληθούν στο πλαίσιο της ΕΦΣΑ. Και αυτή τη στιγμή μας έχουν πει ότι υπάρχει συμμόρφωση με όλους τους κανόνες ασφάλειας των τροφίμων και ότι τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα είναι ασφαλή για ανθρώπινη κατανάλωση. Αυτή είναι η αποστολή της ΕΦΣΑ, αλλά μετά ως πολιτική πρέπει να κάνουμε μια ευρύτερη ηθική συζήτηση. Έτσι πράξαμε και με τα κρέατα που προερχόνται από κλωνοποιημένα ζώα. Και μετά υπήρχε και το ζήτημα φυσικά της εχνηλασιμότητας. Θα πρέπει να μπορούμε να γνωρίζουμε κατά πόσο ένα προϊόν προέρχεται ή όχι από γενετικό τροποποιημένο ε, τρόφιμο ή ζώο. Είναι ε, σχετικά απλό θεωρητικά, αλλά μερικές φορές τα πράγματα περιπλέκονται με τα κλωνοποιημένα ζώα. Διότι οι κλόνοι είναι ακριβώς ταυτόσιμοι γενετικά με τα ζώα από τα οποία κλωνοποιήθηκαν. Μπορούμε λοιπόν να εφαρμόσουμε ένα σωρό κανόνες ασφάλειας ε, και προστασίας ε, αλλά οι απαντήσεις είναι κάτι στο οποίο πρέπει να μας βοηθήσει η ΕΦΣΑ αλλά μαζί με αυτό έχουμε μια άλλη συζήτηση που δεν θα αποφασιστεί από την ΕΦΣΑ αλλά αλλού πρέπει να δούμε πόσο ασφαλή είναι αυτά τα τρόφιμα και πώς μπορούν να αναγνωρίζονται, να γίνεται διάκριση μεταξύ κλωνοποιημένων και μη κλωνοποιημένων τροφίμων. Ευχαριστώ πολύ, Σλούτσερ. Και έχει πάρει τη θέση κυρίας Ρόσπαχ, η οποία είναι τη μεγαλοψυχία της του επιτρέπει. Ναι, ευχαριστώ πολύ γιατί πρέπει να φύγω και πριν από την Λίντα ακόμη. Παρακαλώ λοιπόν ε, τον συνάδελφο να, με παρακολουθ, να παρακολουθήσει απαντήσεις σας. Δεν θα είμαι όμως ο ίδιος παρόν, αλλά επειδή θα μου μεταφέρουν ότι χρειάζεται, θεωρώ ότι δικαιούμαι να αποχωρήσω. Υπάρχει λοιπόν ένα αίτημα για δοκιμές ε, σε μύγες, αυτές που ονομάζονται fruit flies, την κοινή μύγα, ε, στην Ισπανία. Και ίσως σιγά σιγά πάμε και σε μεγαλύτερα ζώα. Δεν καταλαβαίνω όμως γιατί να γίνει τροποποίηση γενετική στα ζώα αυτά, φερειπίν την αγελάδα, εκτός αν, δεν θέλουμε πιο πολύ γάλα, πιο πολύ κρέας, πιο πολύ ανάπτυξη κτηνοτροφίας, δεν καταλαβαίνω ποιος είναι ο λόγος να κάνουμε γενετική τροποποίηση για να βελτιώσουμε την υγεία των ζώων, να αλλάζουμε τα ζώα για να έχουν τι, πιο πολύ χώρο. Όχι. Δεν μπορούμε να κάνουμε ένα ζώο να ε, ωφεληθεί. Δεν, δεν μπορούμε να κάνουμε μια γενετική τροποποίηση από την οποία θα ωφεληθεί το ίδιο το ζώο. Αυτό θέλω να πω. Και επίσης, ε, ξέρουμε ότι οι άνθρωποι δεν θέλουν γενετικά τροποποιημένες τροφές. Άρα λοιπόν, εάν δεν θέλουν οι πολίτες, εάν δεν υπάρχει κέρδος διατροφικό, αν δεν κερδίσουμε σε πιο πολλά προϊόντα, δηλαδή μόνο για να εξυπηρετήσουμε το συμφέρον της εταιρεία που προβαίνει σε αυτήν την, ε, σε αυτήν την ε, τροποποίηση. Και ε, όταν έχουμε μια εταιρεία η οποία τροποποιεί γενετικά τα ζώα της, ε, ωφελείται η ίδια. Εάν όμως πρέπει, επειδή υπάρχει ε, δίπλωμα ευρεσιτεχνία σε ένα γενετικά τροποποιημένο ζώο, ένας κτηνοτρόφος να αγοράζει κάθε χρόνο την πατέντα ή την άδεια εκμετάλλευση του γενετικά τροποποιημένου ζώου, πάλι δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να, να το, επιτρέψουμε αυτό. Είναι ασαφές, αδιαφανές ισχνό το όφελος και αφορά μόνο συγκεκριμένες, συγκεκριμένα συμφέροντα. Δεν έχετε πείσει δηλαδή ότι υπάρχει ανάγκη. Φερρυπίν για την παραγωγή ενός ε, φαρμάκου που θα ήταν χρήσιμο για τον άνθρωπο. Στην ε, παραγωγή τροφίμων δεν βλέπω καμία αιτιολογία που να δικαιολογεί την, ε, κανένα λόγο που να δικαιολογεί την γενετική τροποποίηση. Ερωτώ όμως παρόλα αυτά και επιπλέον Πώς μπορείτε εσείς να εξασφαλίσετε ότι οι μακροπρόθεσμες συνέπειες μίας ιασδήποτε εγκρίσεως, είτε πρόκειται για τη δροσόφυλλο όπως λέγεται αυτή η μήγα, είτε πρόκειται για ένα μεγαλύτερο ζώο, πώς θα το εξασφαλίσετε ότι δεν θα επηρεάσει άλλα ζώα ή φυτά. Πώς έχετε εξασφαλίσει την συνέχεια, το μέλλον και επιπλέον ερωτώ τι είδου συμφέροντα βλέπετε για του πολίτε, για του γεωργού και τι μεγάλε εταιρείε. Όπω είπα, θα χρειαστεί να αποχωρήσω τώρα, αλλά θα ακούσω την απάντησή σα. Θα ενημερωθώ. Ευχαριστώ πολύ. Χάρη στην τεχνολογία, θα τα παρακολουθήσει όλα. Ευχόμαστε και καλή πτήση. Και ακούμε την κυρία Ρόσπαχ και τους υπόλοιπους μετά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αναφερθήκαμε σε μια σειρά κινδυνών. Εγώ θα ήθελα να μιλήσω και για τις πρακτικές πτυχές. Πώς θα μπορούσαμε να εμποδίσουμε τη μόλυνση φυσιολογικών ψαριών από τα, μη, από τα γενετικώς διαπιστώνουμε ότι παρατηρούνται διαρροές ε, στα ενιδρία. Ότι σε εδωτοκαλλιέργειες υπάρχουν διαρροές. Υπάρχουν ε, νούμερα όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο τα γενετικώς τροποποιημένα ψάρια από ηχθειοκαλλιέργειες ε, μεγαλώνουν, ε, είναι πιο, μεγαλώνουν πιο γρήγορα, γίνονται πιο μεγάλα. Ποιο είναι το πλέον έκτημα από την γενετική τροποποίηση. Ήθελα επίσης να μου πείτε πώς ε, η αύξηση των ε, γενετικώς τροποποιημένων επηρεάζει τα ψάρια είπα. Υπάρχει κάποια επισήμενση. Έχουμε πολλά ψάρια από τον Καναδά. Θα πρέπει οι καταναλωτές να γνωρίζουν κατά πόσο αυτά έχουν τροποποιηθεί γενετικά ή όχι. Και επίσης ε, ποιοι είναι οι άλλοι τύποι ζώων σύμφωνα με την ΕΦΣΑ που μπορούν να τροποποιηθούν γενετικά και να βρεθούν στη διατροφική αλυσίδα τα επόμενα χρόνια. Ευχαριστούμε κύριε Λεπάζ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΦΣΑ που ήρθε σήμερα το απόγευμα. Θα συμφωνήσω σε μεγάλο βαθμό με, με τους συναδέλφους, κυρίως με τον Καρ Σλίτερ το πρώτο θέμα είναι η αξιολόγηση και η διαχείριση του κινδύνου. Λοιπόν, να ρωτιόμαστε ε, σε προς τι, σε τι ωφελούν όλα αυτά. Χρειαζόμαστε γενετικά τροποποιημένα ζώα ε, ο στόχος ποιος είναι να ακολουθήσουμε αυτήν την οδό που ακολουθούσαμε με, μια, με ε, έναν τρόπο διατροφής και ένα τρόπο ανατροφής ζών που αντίκειται σε οποιοδήποτε κανόνα ε, ευημερία των ζώων δημιουργούμε, χρειαζόμαστε περισσότερες ζωικές πρωτεΐνες για το σολομό. Εν πάση περιπτώσει, ανεξαρτήτως με το αν θέλουν ή δεν θέλουν οι Ευρωπαίοι αυτά τα ε, ζώα, προς τι. Και νομίζω ότι είναι το βασικό ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί θα είναι επωφελές. Ε, εντάξει, κάποιοι αναρωτιούνται γι' αυτό, αλλά ε, το θέλουμε. Απάντησαν κάποιοι συνάδελφοι ε, με μια σφιγμομέτρη στην Ευρώπη. αν ερωτηθούν οι Ευρωπαίοι αν θέλουν κλωνοποιημένα ζώα, το 98% μάλλον θα πει όχι. Τέλος πάντων, μετά τίθεται το ζήτημα των κινδύνων είναι εξαιρετικά ευρύ αυτό το θέμα, διότι δεν τίθεται το ζήτημα μόνο της υγειονομικής ασφάλειας, δεν είναι ουδέτερο αυτό το θέμα, ε, είναι πάρα πολύ σοβαρό και θα έπρεπε να μελετηθεί μακροχρόνια και εξεπακούεται ότι δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια. Τίθεται όμως και πρόβλημα ε, βιοπικιλομορφίας, ε, γνωρίζουμε ε, τι γίνεται στις υδατοκαλλιέργειες Σολομών, καταλαβαίνετε ότι ότι η φύση δεν λειτουργεί έτσι, θα διαφύγει, ε, θα υπάρξει επιμόλυνση ε, ε, στο υπόλοιπο οικοσύστημα, είναι προφανές. Οπότε θα πρέπει να αναρωτηθούμε με τα έντομα τι θα γίνει, πώς θα επηρεάσουν το υπόλοιπο οικοσύστημα αν μολυνθούν τα έντομα Και διάφοροι χρήστες, ε, άνθρωποι και μη, ε, με ποιο τρόπο θα μολυνθούν από αυτά τα έντομα στη συνέχεια. Ε, κατόπιν το ευζήν των ζώων θα έχουμε μεγαλύτερους σολομούς. Μα δεν είναι φτιαγμένοι γι' αυτό οι σολομοί και το ίδιο ισχύει και για τα υπόλοιπα ζώα. Πέρα είναι ε, το θέμα του κινδύνου, είναι διοντολογικά τα ζητήματα και πέραν αυτό είναι η διαχείριση του κινδύνου που πρέπει ε, να αναλάβουμε εμείς ε, οι πολιτικοί θύνοντες. Είναι δική μας δουλειά και ξαναλέω δεν καταλαβαίνω σε τι βοηθάει. Δηλαδή οι καταναλωτές και πάλι θα έχουν ακόμη μειωμένη, πιο μειωμένη εμπιστοσύνη στην διατροφική αλυσίδα, θα έχουμε ακόμη περισσότερα προβλήματα σε σχέση με αυτά που έχουμε και είναι πολυάριθμα. Ε, νομίζω λοιπόν ότι ε, αυτό είναι το πρωταρχικό ζήτημα. Στο θέσουμε επιτάπητος, ας ε, βγάλουμε τα όπλα που χρειάζεται για να μην επιτρέψουμε να μπουν στην κυκλοφορία αυτά τα προϊόντα που δεν θα προσφέρουν και κανένα όφελος για τους καταναλωτές μας. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Κατίκα παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θα σας εκπλήξει το ότι θα πω ότι δεν είμαι ένθερμη υποστηρικτή των γενετικών τροποποιήσεων και δεν αναφέρομαι μόνο στα ηθικέ πτυχέ του όλου ζητήματο. Τίθεται ένα ερωτηματικό όσον αφορά το περιβάλλον, την βιοπικιλότητα, την υγεία των ζώων καθώ και τη δημόσια υγεία μαζί με πολλούς άλλους συναδέλφους ε, συμφωνούμε ότι ο έλεγχος της διατροφικής αλυσίδας δεν είναι επαρκής. Τώρα μετά τα φυτά μιλάμε για τεχνικές γεννητικές τροπής των ζώων. Έχουμε ελάχιστα στοιχεία για το θέμα αυτό. Ωστόσο, κάποιες πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας δείχνουν ότι με δυσανάλογο τρόπο πολλά ζώα υποφέρουν από αυτές τις διαδικασίες. Η συνθήκη της Λισαβόνα προβλέπει ότι για την υλοποίηση των ευρωπαϊκών πολιτικών πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η καλή μεταχείριση των ζώων. Το απαιτεί όλο και περισσότερο η κοινή γνώμη και κατά την απόψή μου, οι τεχνικέ γενετικής τροποποίησης ε, αντιτίθενται στα όσα προβλέπει η συνθήκη της Λισαβόνα. Αναρωτιέμαι επίσης τι πλεονεκτήματα έχουν όλα αυτά. Υπάρχουν μεγάλα πλεονεκτήματα. Έχουμε κάτι που ονομάζεται προσαρμογή αυτών των ε, τροποποιημένων ζώων που βελτιώνει την αδοχή τους ασθένειες. Εγώ νομίζω ότι θα στα συμπτώματα και όχι στην πηγή του προβλήματος τις εντατικής ε, ε, την κτηνοτροφίας ε, γίνονται προσπάθειες. Πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτό το ζήτημα υπόψη μας των Σολομών που ενδεχομένως θα διαφύγουν και να θέσουμε σε αμφισβήτηση το ζήτημα επίσης της βιοποικιλότητας. Έχω μια ερώτηση προς την ΕΦΣΑ και προς την Κομισιόν. Να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα την για την πολύ ακριβή έκθεση που μας παρουσίασε. Θα μπορούσατε να μας αναφέρετε πώς υπολογίζετε τις μακροχρόνιες επιπτώσεις για το περιβάλλον, την καλή μεταχείριση των ζώων, την δημόσια υγεία. Πώς θα τα εξετάσετε αυτά τα ζητήματα. Θα μπορούσατε επίσης να ε, πραγματοποιήσετε μια μελέτη για να δούμε κατά πόσο υπάρχουν ε, ζώα που αποτελούν το αντικείμενο γενετικής χειραγώγησης θα το ονομαζά έτσι. Πώς θα καταπολεμήσετε τις ε, περιπτώσεις ε, μικροβιακής αντοχής αυτών των ζώων που έχουν τροποποιηθεί γενετικά. Τα ζώα αυτά, τα γενετικώς τροποποιημένα, αποτελούν το αντικείμενο στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων του TTIP. Τι συμπεράσματα έχουν γίνει σε αυτό το θέμα. Η Γενική Διευθυνσή ΣΑΝΚΟ πρόκειται να προσπαθήσει επίσης να παρεμποδίσει και να σταματήσει την Γενική Διευθύνση Εμπορίου, διότι πιστεύω ότι για αυτό το θέμα, για το θέμα της κλωνοποίησης πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γιούζου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλησα να λάβω το λόγο, διότι το μόνο που θέλω είναι να διασφαλίσουμε ότι δεν θα επιβάλλουμε κάτι στους πολίτες, ότι θα μπορούν να το αποφασίσουν ελεύθερα με οποιαδήποτε διασταυρούμενη αναπαραγωγή υπάρχει κάποια χειραγώγηση ουσιαστικά. Μιλάμε τώρα για χειρισμό εντός εργαστηρίου. Ορισμένοι άνθρωποι δίδεται απόλυτα στις γενετικές τροποποίησεις. Τώρα, εάν ένα ανθρώπινο όν γενετικά, μιλάμε για αλλαγές στο γενετικό υλικό, ώστε να δημιουργηθεί κάποια νοσία σε κάποια ασθένεια και τα λοιπά. Τώρα όσον αφορά τη μύγα, υπάρχουν κάποιες γενετικώς τροποιημένες μύγες που δημιουργούνται στο εργαστήριο και μόλις ελευθερωθούν στη φύση ε, συνδυάζονται, αναμεγνύονται με άλλους πληθυσμούς ε, στη φύση που πλήττουν τα φρούτα και με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά η γενετική τροπήση δημιουργεί λιπάσματα κατά κάποιο τρόπο αλλά αυτό που θέλω να ζητήσω από την Εύσα είναι να είναι πολύ αυστηρές οι μελέτες ανεξάρτητες ή όχι, πρέπει να επαληθεύουν ότι διασφαλίζεται η ασφάλεια της ανθρώπινης τροφής, της, ε, των τροφίμων για ανθρώπινη κατανάλωση. Όταν βλέπουμε ένα προϊόν ε, και αναρωτιόμαστε αν ένα γενετικό τροποποιημένο προϊόν είναι κακό για την υγεία των ανθρώπινων όντων, Εάν αυτό έχει αναφέρεται, θα πρέπει να γίνεται σαφές και οι άνθρωποι να μην τρώνε αυτού του είδους το φαγητό. Πρέπει να αποφασίσουμε λοιπόν κατά πόσο τι θα κάνουμε, κατά πόσο μπορούμε, θα μπορούσαμε να, να, να διαθέσουμε ένα εμπόριο γενετικό τροποποιημένο στην αγορά και οι άνθρωποι να αποφασίζουν μόνοι του αν θα το καταναλώσουν ή όχι. Πρέπει να έχουν οι πολίτε την ελευθερία να αποφασίσουν μόνοι του. Εφόσον είναι ασφαλέ, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητής. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και πολύ σύντομα. Μια ερώτηση έχω. Που έχει ήδη διατυπωθεί. Κύριε Τσεξής. Η διατελετική συμφωνία, εταιρική σχέση. Δεν είναι πολύ ο καιρό που είδαμε μια πρόταση εδώ στην Επιτροπή μας για τη χρήση φαλακτικού οξέους για την ε, προετοιμασία, για την επεξεργασία διαφόρων ε, ε, ειδών φερρυπίν σφαγίων ζώων, για επεξεργασία δηλαδή. Και έχω την εξή ερώτηση. Είμαι βιολόγος, τουλάχιστον ήμουν κάποτε βιολόγος δεν διανοούμε να υπάρξουν μέτρα τα οποία μπορεί να οδηγήσουν στον αποκλεισμό της επιμόλυνσης των φυσιολογικών όντων που βρίσκονται στον κόσμο, δηλαδή των μη γενετικά τροποποιημένων από γενετικά τροποποιημένα. Δεν υπάρχει τρόπος να αποκλειστεί η επιμόλυνση. Και μην ξεχνάμε ότι έχουν αναπτυχθεί πολλά ζώα, ε, πολλοί οργανισμοί με μεγάλη αντοχή στα, στους παθογόνους ε, οργανισμούς, στο εγκοπλάσμα πόμπι και άλλους. Και αυτό για μας θα είχε σαν συνέπεια την μια καταστροφή ε, παγκόσμιας κλίμακας για τη δημόσια υγεία. Υπάρχουν επίσης ζώα γενετικά τροποποιημένα στα οποία έχουν εισαχθεί γονίδια που δεν ανήκουν καν στην ομάδα γονιδίων του είδους του ζωικού αυτού. Δηλαδή έχουν προέλθει από άλλους οργανισμούς, από άλλα είδη. Άρα, γιατί η γενετική τροποποίηση μπορείτε να ενισχύσει ένα γονίδιο του υφισταμένου είδους, είτε να εισαγάγει ένα ε, γονίδιο το οποίο δεν ε, ανήκει στον εν λόγω είδος. Εδώ πέρα τι μπορείτε να πείτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να πω ότι έχουμε δύο συναδέλφους από τις μεγαλύτερες ομάδες οι οποίοι συμμετέχουν στην ομάδα TIP και παρακολουθούν την κατάσταση. Ε, ενημερώνουν την Επιτροπή μας τακτικά με, μέσω των συντονιστών και άρα έχουμε παρακολούθηση ως Επιτροπή για το τι συμβαίνει και βέβαια για τα όσα δρομολογούνται. Βεβαίω θα πρέπει να κοιτάξουμε για την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και τι Ευρωπαϊκέ Προδιαγραφέ τι είδου συνέπειε θα φέρει αυτή η Διατλαντική ε, Συμφωνία Εταιρική Σχέση. Θα τα δούμε αυτά. Τα παρακολουθούμε, δεν τα ξεχνάμε. Κύριε Πουλέ ή κάποιος άλλος. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Si vous... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα ε, να αρχίσω ε, απαντώντας και μετά η, η θα απαντήσει στα ερωτήματα που απίφθηναν ε, τα μέλη της Επιτροπής ε, στον ΕΦΣΑ. Ε, θα ταξινομήσω τις απαντήσεις σε πέντε κατηγορίες, αν μου το επιτρέπετε. Πρώτον, ναι, ποια είναι τα υποτιθέμενα ωφέλη. Ο Σολομός, ε, όπως παρουσιάστηκε η περίπτωση στη ΣΥΠΑ, αλλά θα καταλάβατε ότι δεν εκτρέφεται στη ΣΥΠΑ, ε, τα έμβρια του Σολομού παράγονται στον Καναδά και τα ενήλικα ψάρια στον Παναμά. Ο στόχος είναι να να αυξάνει το πάρος του με διπλάσιο ρυθμό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, δεν είναι σε θέση να σας πει ότι θα μειωθεί δύο φορές και η τιμή του αντίστοιχα. Ε, δεν ξέρουμε τίποτα γιατί προς το παρόν δεν κυκλοφορεί στην αγορά. Αλλά πάντως αυξάνει το βάρος του ε, με διπλάσιο ρυθμό με την ίδια ποσότητα ζωοτροφής. Οπότε μπορεί κανείς να υποθέσει ότι υπάρχει οικονομικό όφελος για τις εταιρείε που θα αναλάβουν την εκτροφή. Όμως δεν μπορώ να σας πω περισσότερα πράγματα γιατί δεν ξέρουμε κιόλας. Για τα υπόλοιπα ζώα ε, αληθεύει ότι υπάρχει περίφημη αυτή τροσόφιλος ε, μίγα και έχει, υπάρχει ένα ισπανικό ερευνητικό πρόγραμμα. Είναι παθογόνος αυτή ε, η μίγα. για την ελιά και ξέρετε ότι ε, υπάρχουν διάφορα σενικά έντομα που βομβαρδίζονται ραδιενεργώς με κοβάλτιο για να μην αναπαράγονται και ε, απελευθερώνονται στη φύση, βρίσκουν ένα, ε, ένα θηλυκό ε, την ε, γονιμοποιούν, όμως ε, δεν υπάρχουν γονιμοποιημένα οάρια λόγω της ραδιενέργειας και δεν αναπαραγονται, πολλαπλασιάζονται έντομα. Εδώ και 30-40 χρόνια υπάρχουν αυτά τα προγράμματα και χρησιμοποιούνται ραδιενεργές ουσίες για αυτή τη δροσόφυλλο λοιπόν το ζήτημα είναι να ε, τροποποιηθεί γενετικά για να είναι στήρο το αρσενικό έντομο και άρα να μην γονιμοποιηθούν τα οάρια ε, του θηλυκού εντόμου και εφόσον το θηλυκό μπορεί να γονιμοποιηθεί από ένα αρσενικό δεν ε, υπάρχουν Ε, δεν αναπαράγεται. Ε, οπότε ε, υπάρχει και το άλλο το ζήτημα τώρα με τα εντομοκτώνα, τα παρασιτοκτώνα. Υπάρχουν ε, ε, δοκιμές ε, σε πραγματική κλίμακα στην Ισπανία ή τουλάχιστον σχεδιάζονται για να δούμε αν υπάρχουν οικονομικά ωφέλη για τις νέες τεχνικές για τα βορειοστοκτόνα και πρέπει να δούμε όμως αν αυτά που γίνονται για τις, τις μύγες επηρεάζουν τις μύγες ή άλλα έντομα αρνητικά προτού προχωρήσουν αυτά τα ερευνητικά προγράμματα. Υπάρχουν και βακτήρια που τροποποιούνται γενετικά ούτως ώστε να ε, παράγουν φαρμακευτικά σκευάσματα στη συνέχεια δεν είναι όμως αμφιλεγόμενο το ζήτημα, διότι τα φαρμακευτικά σκευάσματα χρησιμοποιούνται για την ίαση των ανθρώπων ε, και ε, ο στόχος είναι αναπαραγωγή ορμονών όπως η ινσουλίνη. Χάρη σε αυτά τα ε, βακτήρια, αντί να παίρνουμε από τα σφαγεία ορμόνες από τα ζώα που ενδεχομένως έχουν μολυνθεί. Αυτό δεν είναι αμφιλεγόμενο ζήτημα. Ξέρουμε επίσης ότι υπάρχουν έρευνες για ε, τους χείρους για να ε, ανθίστανται ε, στην γρήπη των χείρων ε, ή σε άλλες, ε, ε, σε νόσους. Υπάρχουν και τα αγριογούρουνα που προσβάλλονται από αυτές τις νόσους. Βεβαίως δεν εκτρέφονται με εντατικό τρόπο όπως οι Στο στάδιο το τωρινό πάντως οι έρευνες προχωρούν και δεν υπάρχει αμφισβήτηση. Δεύτερο ζήτημα, δεοντολογικά ζητήματα. Ο κανονισμός Οδηγία 2001, Κανονισμός 2009. Υπάρχουν διάφορα ζητήματα που μπορούμε να θέσουμε για να δώσουμε απαντήσεις σε αυτά τα διοντολογικά ε, ερωτήματα. Προσοχή όμως όταν ε, χειριζόμαστε τα ζητήματα διοντολογίας ε, μετά από την παρουσίαση του προγράμματος δεν αποκλείουμε το ενδεχόμενο να ζητήσουμε γνωμοδότηση από την Ευρωπαϊκή Διοντολογική Επιτροπή που έχει ήδη εκδώσει ε, γνωμοδότηση το 96 συγκεκριμένα, για τις ε, ε, φυσιολογικές τεχνικές, τεχνικές συγγνώμη, γενετικά τροποποιημένων ζώων. Πρόκειται για ζώο, περίφημος αυτός ο λομός, και ε, το κρέας του ε, προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση. Δεν αποκλείεται να ε, ζητήσουμε να εκδώσει εκ νέου γνωμοδότηση η Επιτροπή Διοντολογίας. Τρίτη κατηγορία, κίνδυνη. Για, η κίνδυνη για την δημόσια υγεία είναι προφανές, η ΕΦΣΑ ασχολείται με αυτό, κίνδυνος για το περιβάλλον, Επίσης ε, θα αξιολογηθεί από τον ΕΦΣΑ ε, επίπτωση επί της βιοπικιλότητας πάλι θέμα του, της Ευρωπαϊκής Αρχής ε, Τροφίμων. Υπάρχει όμως το ζήτημα του εγκλισμού αυτών των ζώων. για τα ψάρια στο Παναμά, για τους ολομούς στο Παναμά, ε, επευλήθη να μην εκτρέφονται στην ε, ανοιχτή θάλασσα αλλά σε δεξαμενές ε, περίκλειστες Ξέρετε ότι όταν η κλωβή είναι στην ανοιχτή θάλασσα λόγω των ε, οπών που μπορεί να υπάρχουν ε, στα δίχτυα στους κλοβούς, μπορούν να διαφύγουν οι σολομοί και να αναπαραχθούν με ε, άγριους σολομούς και το καθεξής. Για να αποφευθεί αυτός ο κίνδυνος και η επιμόλυνση των αγρίων ειδών οι Αμερικανοί αποφάσισαν να εκτρέφουν ε, τα ε, ψάρια, όπως σας είπα, σε τους κλοβούς με ε, φίλτρα που καθαρίζουν το νερό που χρησιμοποιείται κατά την απορροή του, ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος επιμόλυνσης. Χερσαία λοιπόν εκτροφή η σολομή, η ε, σε παραδοσιακή ή γενετικά τροποποιημένη ε, πρέπει να συμμορφώνονται ε, ως προς την εκτροφή τους εννοώ με κάποια μέτρα για το ευζήν των ζώων εάν ήταν δυνατή, και το τονίζω εάν ήταν δυνατή η εκτροφή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα υπήρχε συμμόρφωση με αυτέ τι απαιτήσει. ε, τέταρτη κατηγορία, συμφέροντα του καταναλωτή. Ε, Όντω ε, υπάρχει μια πολιτική επιλογή που πρωτίστω πρέπει να γίνει. Η Επιτροπή ε, και ο Επίτροπο το τόνισε, ούτε υπέρ ούτε κατά είναι. Εφαρμόζει τον κανονισμό που προετοίμασε και εξέδωσε το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Ε, η απαγόρευση συνιστά πολιτική επιλογή. Εάν αυτά τα δύο θεσμικά όργανα αποφάσιζαν την πλήρη απαγόρευση των γενετικά τροποποιημένων ζώων, είναι προφανές ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εφαρμόσει την απόφαση αυτή. Προς το παρόν, ρυθμίζονται αυτά τα ζητήματα, όπως σας ε, είπα, ε, από την οδηγία και τον κανονισμό, όπου δεν απαγορεύεται ένα γενετικά τροποποιημένο ε, ζώο, όμως υποβάλλεται σε απαιτήσει σήμανσης για να ενημερωθεί ο καταναλωτής και οποιοδήποτε προϊόν παράγεται από αυτό το ζώο. Επίσης υπάγεται στην υποχρέωση σήμανση, όχι μόνο το κρέας του σολομού, αλλά και το λάδι, τα ηχθιάλευρα που χρησιμοποιούνται για τις ζωοτροφές, για την κτηνοτροφία, και ούτω καθεξής. Όλα αυτά ε, υπάγονται στην υποχρέωση σήμανσης όπως και τα προϊόντα φυτικής προελεύσεως με τρόπο ώστε ο καταναλωτής να μπορέσει εν πλήρη συνειδήση να κάνει τις επιλογές του και να καταναλώσει ή όχι. Πέμπτη κατηγορία. Σχέσεις ε, με τη ΣΥΠΑ στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία TTIP. Ο πρόεδρος Μπαρόσο ήταν ξεκάθαρος ε, όταν ξεκίνησε κίνησαν αυτές οι διαπραγματεύσεις ε, πριν από λίγους μήνες ε, δεν τίθεται ζήτημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη ΣΥΠΑ να συζητήσουν για το ενωσιακό επίπεδο προστασίας ε, ως προς τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Είναι προφανές ότι ανταλλάσσουμε επιστημονικές πληροφορίες σε σχέση με την αξιολόγηση του ΕΦΣΑ, σε σχέση με τη διαδικασία έγκρισης, το τι εγκρίνουμε, τι δεν εγκρίνουμε κτλ όμως δεν τίθεται ζήτημα διαπραγμάτευσης ε, τροποποίησης ε, του κανονισμού, αυτή η περίφημη οδηγία που σας έλεγα προηγουμένως και ο περίφημος κανονισμός, ε, στα πλαίσια της TTIP. Είναι ταμπού στις συζητήσεις που γίνονται για την διαπραγμάτευση της TTIP. Παρότι, όπως σας είπα, γίνονται συζητήσεις και είπα μας ρώτανε γιατί χρειάζεται μία πενταετία ως και δεκαετία για να εγκρίνεται ένα γενετικά τροποποιημένο ενώ εμείς χρειαζόμαστε ένα χρόνο. Πέραν αυτού τους εξηγούμε τις διαδικασίες που ακολουθεί ο ΕΦΣΑ, τις πολιτικές, ε, τα πολιτικά κολλήματα κτλ. Αλλά πέραν αυτού ε, δεν τίθεται ζήτημα να αρχίσουμε να συζητούμε μαζί τους την τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας. Ιδού, Πρόεδρε, εγώ αυτά ε, μπορούσα να απαντήσω από πλευράς της Επιτροπής ε, και τώρα η συνάδελφος από τον ΕΦΣΑ θα δώσει πιο τεχνικές απαντήσεις. Ευχαριστούμε κύριε Πουλέ. Θα δώσουμε στην κυρία Μπέγμαν αμέσως τον λόγο να μας απαντήσει εξ ονόματος του ΕΦΣΑ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι σίγουρα δεν έχουμε καμία αρμοδιότητα για τα πλεονεκτήματα, αλλά έχουμε αρμοδιότητα για να ελεγξούμε την περιβαλλοντική ασφάλεια και ένα από τα δύο έγγραφα που εκπονήσαμε αφορά ακριβώς αυτό το ζήτημα. Τα δύο έγγραφα που τελούν κατευθυντήρες γραμμές. Αυτό σημαίνει ότι κάνουμε ερωτήσεις. Έχουμε ένα κατάλογο ερωτήσεων και παρέχουμε κάποιες κατευθυντήριες γραμμές για την δημιουργία στοιχεία για τον ετούντα, ώστε να δημιουργηθεί ένα πακέτο στοιχείων. Με αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές δεν απαντάμε ακόμα τις ερωτήσεις, διότι πρώτα πρέπει να λάβουμε το σύνολο των δεδομένων για να το κάνουμε αυτό. Εσείς κάνετε πολλές ερωτήσεις που θα έπρεπε να σε απαντήσει ο ετών με τα δικά του στοιχεία, τα οποία θα πρέπει να καταρτήσει ο ίδιος. Ρωτήσατε τι γίνεται αν διαφύγει ένα γενετικό τροποποιημένο ψάρι, τι γίνεται με το περιβάλλον, τι συμβαίνει με τους άλλους πληθυσμούς ψαριών. Είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να σε απαντήσει ο ετών. Επίσης άκουσα μια ερώτηση που τι γίνεται με τους ε, ανθρώπους, τι συμβαίνει σε αυτούς αν έρθω σε επαφή με ένα γενετικό τροποποιημένο έντοπο το ίδιο ετών πρέπει να απαντήσει. επίση ποιε είναι οι συνέπειες όσον αφορά την αντοχή σας ασθενή στην ανοσία σε θέματα ευημερία των ζώων. Και αυτό πάλι το απαντά ένας ετών. Δεν μπορώ εγώ λοιπόν να σα το απαντήσω, αλλά ο ΕΦΣΑ ζητά στοιχεία για να ψάξει να βρει ποιε θα ήταν οι απαντήσει σε περίπτωση που ένα τέτοιο ζώο κυκλοφορεί στην αγορά. Από αυτή την έννοια θεωρώ ότι ήμασταν ιδιαίτερα επιμελείς. Έχουμε πέντε διαφορετικές ομάδες εργασίας ώστε να μπορέσουμε να διαπιστώσουμε ποιες είναι οι σωστές ερωτήσεις. Και φυσικά η αρχή της κατά περίπτωση εξετάσεις είναι πολύ σημαντική γιατί ανάλογα με το ζώο που έχουμε μπροστά μας, ανάλογα με το τι είδου γενετική τροπή έχει υποστεί, χρειάζεται κανείς να εστιαστεί σε διαφορετικές ερωτήσεις. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στη συναδελφό μου, Σιλβί Μέστακ, η οποία ήταν επιφορτισμένη με το έγγραφο αξιολόγησης ε, περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπου εξετάστηκαν τρεις τύποι ζώων με τρεις διαφορετικούς τύπους γενετικών τροποποιήσεων. Ευχαριστώ, Σίλβη. Yeah, bitte. Ευχαριστώ πολύ. Yeah, thank you. Σας ευχαριστώ. Θα θέλω να αναφερθώ στις ε, κατευθύνσεις που ανέπτυξε ο ΕΑΤ, η ΕΦΣΑ πρόσφατα, και να συνδέσω με δύο σημαντικά θέματα. Καταρχάς η αξιολόγηση πιθανών μακροπρόθεσμων συνεπειών και πιθανολόγηση ή πιθανότητες διαφυγής στη φύση ενός γενετικά τροποποιημένου ζώου μακροπρόθεσμο συνέπειες βεβαίως μπορούμε να αξιολογήσουμε μόνο με βάση τα όσα γνωρίζουμε κατά τη στιγμή της αξιολόγησης ασφάλειας. Δηλαδή ε, ζητούμε από τον ετούντα και από τον αξιολογούντα γενικά τον κίνδυνο να προσφέρει τις βέλτιστες δυνατές ή τις πλήστες όσες πληροφορίες για κάθε τι, πειραματικά στοιχεία, ε, χρήση με τα ζώα υποκατάσταση όπω ονομάζονται, δηλαδή αυτά που έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά αλλά δεν είναι γενετικά τροποποιημένα, γιατί αυτό μπορεί να μας διαφωτίσει και αναλόγως στοιχεία τα οποία μπορούν να μας ε, βοηθήσουν σε μακροπρόθεσμες ε, ε, αξιολογήσεις. Και βέβαια έχουμε και την, και την παρακολούθηση στην περίοδο μετά τη διάθεση στην αγορά όπως ισχύει για τα φυτά, η μεθοδολογία είναι ίδια και για τα ζώα. Στόχος μας είναι, τώρα όπως λέτε με την ερώτηση για το αν υπάρχει κίνδυνος να διαφύγει ζώο στη φύση, ε, βεβαίως είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να εξετάσουμε. Τα νέα χαρακτηριστικά του ζώου μπορεί να Ε, μπορούμε να τα παρακολουθήσουμε, μπορούμε να δούμε τι είδους συνέπειες μπορούν να έχουν. Ε, όλα αυτά τα ζητάμε από την επιχείρηση, από την εταιρεία που έχει αναπτύξει τον γενετικά τροποποιημένο οργανισμό να μας τα δώσει. Λίγο πολύ αυτά. Απλώς για να ολοκληρώσω κατά την αξιολόγηση κινδύνου. Αφού έχουμε, τον, ε, αφού έχουμε χαρακτηρίσει τον κίνδυνο, προβαίνουμε και σε μια αξιολόγηση των μέτρων μετριασμού του κινδύνου που θα μπορούσαμε να έχουμε και βέβαια ανάλογα εκτιμούμε αν χρειάζεται να προτείνουμε, αν είναι χρήσιμο. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Είχε, νομίζω, άξιζε τον κόπο να δώσουμε αυτό το χρόνο και να το συζητήσουμε. Έστω και αν πέμπτη απόγευμα Πολλοί έχουν, έχουν επανέλθει στις αιστείες τους, ε, στις εκλογικές τους περιφέρειες, είμαστε ίσως ολιγάριθμοι, αλλά πάντως όσοι άντεξαν ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ πολύ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον ΕΑΤ, όλους τους συναδέλφους που είναι εδώ για τη συζήτηση και έτσι νομίζω ότι ε, εξαντλήσαμε την ημερησία μας διάταξη. Θα τα ξαναπούμε μαζί με την Επιτροπή Ήτρε για τους, στίχους, για τους στόχους 2030 2 Δεκεμβρίου. 3 με 6 το απόγευμα, 3 με 6,5 το απόγευμα και 16-17 Δεκεμβρίου πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων. Ακρόαση. Σημειώνετε παρακαλώ και καλό σας βράδυ.